Ladies and gentlemen, please be... Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Καλημέρα σας. proszę Państwa, zaczynamy. Άρχεται η συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Και καλωσορίζω θερμότατα τα μέλη της Υποεπιτροπής και τους καλεσμένους μας. και τους συμβούλους Φυσικά καλωσορίζω θερμότατα τον πρώτο μας καλεσμένο, τον πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον στρατηγό Πατρίκ Ντερουζιέ. Επιτρέψτε μου κύριε στρατηγέ, στρατηγέ μου, να υπενθυμίσω την, την ε, ημερήσια διάταξη. Καταρχήν να σας ενημερώσω ότι έχουμε διερμηνία για τα τακτικά μέλη της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Προηγούνται στη διερμηνία τα τακτικά μέλη. Επίσης, η συνεδρίασή μας μεταδίδεται απευθείας στο διαδίκτυο. Υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Την έχετε λάβει από τη γραμματεία, παρακαλώ. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω τον στρατηγό Πατρίκ Ντερουζιέ που επαναλαμβάνω είναι πρόεδρος της ε, Στρατητικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η Στρατητική Επιτροπή είναι το ύπατο συμβουλευτικό όργανο για στρατητικά θέματα του Συμβουλίου και έχει αρμοδιότητα να παρακολουθεί και να φροντίζει για τη σωστή εκτέλεση των, Ευρω... των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι βεβαία ότι επειδή έχουμε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και πολλές απειλές στην κοινή μας ασφάλεια, και αντίθετα με τις ε, διατάξεις της ε, στρατηγικής μας για την ασφάλεια του 2003, Και ακριβώς επειδή έχουμε απειλές ασφάλειας σε άμεσα γειτονικέ χώρες και επειδή έχουμε πραγματική πυρκαγιά στα σύνορά μας και προς Ανατολάς στην Ουκρανία αλλά και άλλο στη Βόρεια Αφρική για παράδειγμα στη Μέση Ανατολή η κατάσταση είναι φλέγουσα. Σήμερα λοιπόν θα εξετάσουμε και τις προκλήσεις στη Συρία και το Ιράκ και την απειλή που δημιουργεί η οργάνωση Ισλαμικό κράτος. Στρατηγέ μου, φαντάζομαι θα σχολιάσετε αυτά τα θέματα στην ομιλία σας και θα μας εκθέσετε και τις δικές σας απόψεις για τις τρέχουσες αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ικανότητά μας να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τους μηχανισμούς και τα μέσα που έχουμε με βάση τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Στρατηγιά μου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι και τιμή και χαρά για μένα να παρίστα με εδώ και να μπορώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας για τις στρατιωτικές διαστάσεις των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είχα την ευκαιρία να αναφέρω πρόσφατα, κατά τη διάρκεια των δύο ετών στη θητεία αυτή, η ανταλλαγή απόψεων αποτελεί μια προνομιούχα στιγμή, ε, της οποίας τη σπουδαιότητα κατανοώ απόλυτα. Από το Σαχέλ μέχρι το Ιράκ, την Ουκρανία μέχρι τη Συρία ή την Λιβύη, αλλά και εκτενέστερα με την διάδοση του ιού έμπολα, η βαρύτητα, ο σύνθετος χαρακτήρας και η έκταση των κρίσεων που αντιμετωπίζουμε αντιπροσωπεύουν πιθανούς, ισχυρούς πιθανούς κινδύνους αστάθειας στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Υπήρου αλλά και πέραν της ε, κοντινής γειτονιάς μας θέτουν και μας υποχρεώνουν να επανεξετάσουμε την προσέγγιση μας για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Γι' αυτό ως πρόεδρος της, Επιτροπής, της Στρατιωτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω καταρχά να μιλήσω ενώπιον σας για τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι, τον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα θεωρούνται από τις διάφορες, ε, από των στρατιωτικών δυνάμεων των στρατών στην Ευρώπη και τους οποίους εκπροσωπώ. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι τι μπορούμε να κάνουμε και τι απαντήσεις προσπαθούμε να δώσουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας. Ξεκινώ από την άποψη των επικεφαλής των επιτελείων για την διεθνή κατάσταση. Η ανάλυση που κάνουμε είναι ότι οι απειλές που αντιμετωπίζουμε ξεπερνούν κατά πολύ το πλαίσιο των κρατών. Ενισχύουν ταυτόχρονα και την άποψη για την ανάγκη να να διευρυνθεί η αμυντική δράση προστασία συνόρων και του πληθυσμού. Υπάρχει μια αντίφαση λοιπόν μεταξύ της βασικής δράσης των στρατιωτικών προστασία του εδάφους από κάθε ένοπλη δύναμη σε κάθε χώρα και αφετέρου από την έννοια ότι μόνο μόνοι μας δεν μπορούμε να δράσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Η, κατάσταση, η διεθνής αυτή κατάσταση αφορά πρώτον την κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη που ταράσει την αρχή του απαραβίαστου των συνόρων και οδηγεί στο να επανεξετάσουμε, να ξαναδούμε την έννοια της ελεγγύης μεταξύ Ευρωπαίων. Ένα άλλο θέμα είναι ο διεθνής, η διεθνής τρομοκρατία που δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ καλά μπορεί να χτυπήσει στην καρδιά των κοινωνιών μας, των ε, χωρών εταίρων αλλά και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στο εξωτερικό. Πρόκειται επίσης για το οργανωμένο έγκλημα διακίνηση ατόμων, όπλων, ναρκωτικών που δημιουργούν ζώνες αναταραχής σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην Αφρική, σε έναν άξονα κρίσεων που ξεκινάει από τις ακτές του Ατλαντικού μέχρι τον Ινδικό ωκεανό. Πρόκειται για την πειρατεία, την ληστεία των θαλασσών που αντιπροσωπεύουν πάντα μια απειλή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε γιατί ε, φύγει τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης φέτοντας σε κίνδυνο τις ροές ε, τροφοδοσίας της Ευρώπης θέλω επίσης να θυμίσω, πρόκειται και για το κυβερνοχώρο που αντιμετωπίζει τακτικές επιθέσεις και των οποίων αναπτύσσουμε συστήματα προειδοποίησης και πρόληψης που επιτρέπουν την, το να μοιραζόμαστε πληροφορίες αλλά και προφανώς αυτό είναι ε, ένας χώρος όπου οι στρατιωτικοί μπορούν να συμβάλλουν κάπως την αντοχή, την ανθεκτικότητα. Με αυτό το γρήγορο πανόραμα κρίσεων, πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις απειλές, αυτές τις κρίσεις. Σήμερα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις που είναι αποτελεσματικές, καινοτόμες, ικανές να συμβάλλουν στην διεθνή σταθερότητα αλλά και στην ασφάλεια του, της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Όπως γνωρίζετε, στα πλαίσια της ΕΠΑ, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλισης, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε δυνατότητα να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά εργαλεία, περιορισμένα βέβαια, αλλά κάθε μέρα αυτό το στρατιωτικό εργαλείο αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του. Δεν δρά μόνο του. Είναι σημαντικό διότι είναι συμπληρωματικό άλλων δράσεων που διεξάγονται προς ε, όφελος των συνολικών πολιτικών που επιθυμούν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συντονισμένη, όπω αποκαλούσα προσέγγιση, είναι ένα ουσιαστικό ατού γιατί επιτρέπει στην Ένωση να μην περιοριστεί στις αντιδράσει όταν αναδεικνύονται οι κρίσει, αλλά να προλάβει, να προεξοφλήσει και να προσπαθήσει να τις, λύσεις, να τις λύσει μόνιμα. Ωστόσο, ε, καλό θα ήταν να θυμίζουμε ότι δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκό στρατός με την κλασική έννοια του όρου. Η άμυνα της Ευρώπης διασφαλίζεται πάντα από το κάθε κράτος μέλος που ατομικά έχουν τον έλεγχο των αμυντικών δομών τους και την υλοποίηση των, ε, της, του δυναμικού τους. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο των ε, Υπουργείων Αμήνης κάθε χώρας. Επιπλέον, συνολικά, σε ό,τι αφορά τη συλλογική άμυνα, το ΝΑΤΟ είναι αυτό που έχει την βασική ευθύνη. Η Ευρώπη της άμυνας λοιπόν δεν είναι μια, Ευρώπη, μια άμυνα κλασικής, αλλά μια πολυεθνική φιλοδοξία, μια αλληλεγγύη κυρίω που εκφράζεται με, ανάλογα με τις κρίσεις και τη βούληση εμπλοκής των 28 κρατών μελών. Για μένα η Ευρώπη της άμυνας είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Πράγματι, σήμερα έχει παρέλθει ο χρόνος της στρατηγικής απομόνωσης. Σε αυτή, γιατί για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, συχνά υπάρχει τάση να αντιδρούμε σε ατομικό και ανεξάρτητο επίπεδο για λόγους ευελιξίας. Σήμερα ωστόσο συμπληρωματικότητα είναι υποχρεωτική επιταγή γιατί προσφέρει και, παρα, και κατανομή πολιτικής ευθύνης, εγγύηση αλληλέγγυας δέσμευσης και, κάτι εξίσου σημαντικό, δέσμευση στο χρόνο. Αυτή η συμπληρωματικότητα μπορεί να ασκηθεί σε κάθε επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο εμπλοκής, αλλά και στη φάση της προετοιμασίας. Μπορεί λοιπόν να ε, λειτουργήσει με διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, διμερός. Για παράδειγμα, αυτό είναι η συνεργασία των πεζοναυτών Βελγίου και Ολλανδίας που ενοποίησαν τους στόλους τους για να υπάρξει ένα διεθνές, διεθνικό στρατηγείο που βρίσκεται στην Ολλανδία. Το ίδιο ισχύει και όταν υπάρχουν ομαδοποιήσεις συμφερόντων για παράδειγμα στην περίπτωση του φόρουμ Νορντεύκο, μέσα στο οποίο η Δανία, η Φιλανδία και η Σουηδία μετέχουν μαζί με την Ισλανδία και την Ορβηγία σε κοινέ ασκήσει ετοιμάζουν ε, κοινά πλαίσια διαχείριση κρίσεων και συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της ομάδας του Βίσεγκρατ μεταξύ Τσεχίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας και Σλοβακίας που πρόσφατα αποφάσισαν να προσεγγίσουν στον τομέα τη συνεργασία και του προγραμματισμού της άμυνας. Το ίδιο γίνεται και στη συνεργασία με διεθνείς φορείς. Για παράδειγμα, στο Σαχέλ υπάρχει μόνιμος διάλογος με περιφερειακούς ε, δρόντες, ιδίως το σύστημα ενημέρωσης της αστυνομίας της Δυτικής Αφρικής, το πρόγραμμα δράσης του ΣΕΝΤΕΑΟ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και, την, και της εγκληματικότητας και βεβαίως την Αφρικανική Ένωση. Αφετέρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ε, το επιβάλλει λογική, συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ. Η εμπλοκή των κρατών μελών στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας είναι και θετική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει και για την επεξεργασία κοινών ε, δυνατοτήτων, αλλά και για την κατανομή των ευθυνών, όπως βλέπουμε ε, στην Αφρική και στο Σαχέλ και στο κέρας της Αφρικής. Η δυναμική αυτή μπορεί να μόνο να διευρυνθεί μπορεί στο μέλλον, γιατί η, απάντηση, η απόφαση των αρχηγών κρατών κυβερνήσεων στο Νιούπορτ μας το επιβάλλουν. Πρέπει κατά συνέπεια να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε να προχωρούμε και να εντατικοποιούμε τον, την πορεία αυτή, ούτω ώστε οι συνεργασίε μεταξύ Ατλαντική Συμμαχία και Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδεθούν περισσότερο. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Αλλά να ξαναμιλήσω τώρα λίγο για τι επιχειρησιακέ παρεμβάσει μα. Σήμερα, όπω ξέρετε, η Ένωση έχει ταυτόχρονα πέντε επιχειρήσει, στρατιωτικέ επιχειρήσει, κάτι που ήταν ανήκουστο. 3.000 στρατιώτε στρατιώτες από τις χώρες Ευρώπης αυτή τη, στιγμή, τη στιγμή βρίσκονται κάτω από την Ευρωπαϊκή Σημαία και διαφοροποιούν την κατάσταση. Αυτοί, χάρη σε ισχυρές εντολές, συμβάλλουν καθοριστικά στην ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια. Είναι αποστολές συμβουλευτικές και αποστολές υποστήριξης για τη μεταρρύθμιση της ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα και ειρηνευτικές επεμβάσεις και δια... και, και, και βοήθεια στην επίλυση κρίσεων. Τώρα, τι γίνεται με τις διάφορες περιπτώσεις. Θα αναφερθώ μία προς μία. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Όπως ξέρετε, τον περασμένο Φεβρουάριο ο Ιωάννης ξεκίνησε τη στρατιωτική επιχείρηση U4RCA με στόχο να δημιουργηθεί προσωρινά ένα ασφαλές περιβάλλον στην περιοχή του Μπαγκούι και να συμβάλλει στις προσπάθειες για να προστατευτεί ο πληθυσμός εκεί και να διευκολυνθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε σε πλήρη δυναμικό η δύναμη και αυτή τη στιγμή εξασφαλίζει την ασφάλεια του αεροδρομίου του Μπαγκούι, λειτουργεί αυτό δηλαδή, και επιπλέον ε, έχει επεκταθεί και στο τρίτο και πέμπτο τομέα της πόλης. Σήμερα 750 στρατιώτες και χωροφύλακες της επιχείρησης αυτής δραστηριοποιούνται στο Μπαγκούι και με αποτελεσματικό τρόπο συνέβαλαν στη μείωση του επίπεδου ασφάλειας. Κάποια παραδείγματα. Το προσωπικό που μετακινείται στο εσωτερικό, δίπλα στο δρόμιο ξεκίνησε να επιστρέφει στον τρίτο και πέμπτο τομέα. Όταν φτάσαμε υπήρχαν 100.000 διωγμένα άτομα. Πολλοί είναι και τώρα, αλλά μόνο 20.000 πια. Κάποιοι κεντροαφρικανοί είχαν διαφυγή στο Τσάντ. 3.000 από αυτούς επανήλθαν στις περιοχές αυτές. Αυτή η συλλογική επιτυχία στηρίζεται στην, στην εμπλοκή όλων. Μεταξύ της ιδιαιτερότητας αποστολής αυτής είναι ότι για πρώτη φορά δίπλα-δίπλα σε συνέργεια υπάρχουν στρατιώτες και χωροφύλακες. Πρόκειται για μια συντονισμένη προσέγγιση που επιτρέπει να διευκολύνουμε δράσεις εμπλοκής και του πληθυσμού. Η ίδια επιτυχία περιλαμβάνει και την εμπλοκή των ντόπιων και ντοθεκανικών δυνάμεων που κάνουν κοινέ επιχειρήσεις με τους Ευρωπαίους χωροφύλακες αλλά που ε, και που συνεργάζονται και με την Μίσκα και εδώ και λίγο καιρό με την Μίνουσκα. Όπως γνωρίζετε, για να ενθαρρύνουμε μια ε, αποτελεσματική μετάπτωση, ε, συνεργασία μεταξύ των, της δικής μας αποστολής και της αποστολής του ΟΗΕ, μελετάμε μια μικρή παράταση της αποστολής μας που θα μπορούσε να επεκταθεί μέχρι το Μάρτιο του 2015. Έχουν ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις και αναμένεται μια πολιτική απόφαση τις επόμενες εβδομάδες. Δεύτερος τομέας δράσεων η γνωστή επιχείρηση EUNAFOR Atalanti, πολέμηση της πειρατείας, που είναι πάντα χρήσιμη και αποτελεί σημείο αναφορά στην περιοχή για δράσεις κατά της πειρατείας και που από το ξεκίνημά της, το τέλος του 2008, επέτρεψε στο Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα να διανύει 960.000 τόνους τροφίμων στην περιοχή και μάλιστα με ασφαλή τρόπο είναι πραγματικά σημείο αναφορά στην περιοχή αυτή. Γι' αυτό και έχουμε ε, και από εξωτερικού παράγοντε προσκλήσει για συνεργασία από την Ιαπωνία, την Κίνα, τη Νέα Ζηλανδία και ε, πολλέ άλλε χώρε. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τις ε, διάφορες εναλλακτικές λύσεις για το μέλλον, πώς και αν χρειάζεται να τροποποιήσουμε την επιχείρηση αυτή. Θα πρέπει όμως να έχουμε κατά νου την ανάγκη επαγρύπνησης και εγρήγορσης για να αντιμετωπίσουμε απροσδόκητες καταστάσεις και φυσικά το σημαντικό έργο που είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για να διατηρήσουμε τις δράσεις μας. Τώρα, η επιχείρηση ε- EU4 Altea στα Βαλκάνια που συμβάλλει στην σταθερότητα και την εξασφάλιση της, και την προστασία της ασφάλειας στη Βοσνία και Ζεγοβίνη. Οι πλημμύρες του Μαΐου επιδίνωσαν την οικονομική κατάσταση της χώρας και έδειξαν ότι ε, έχει καταστεί πιο έθραυστος ο δεσμός μεταξύ του πληθυσμού και των πολιτικών εθνών. Και μάλιστα η παρουσία των στρατιωτικών, της στρατιωτικής δύναμης Αλτέα συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο στη διατήρηση της ασφάλειας. Βέβαια, οι στρατιώτες συνεχίζουν τις, την αποστολή εκπαίδευσης, βοηθώντας τους στρατιωτικούς της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και συμβάλλουν στις διάφορες επιχειρήσεις που γίνεται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Τέλος, τρίτος πυλώνας των δράσεών μας είναι η συμβολή μας ώστε να μειωθεί ε, το πλωστάσιο ε, και τα πυρομαχικά στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ε, είναι υπερβολικός ο αριθμός των όπλων και των πυρομαχικών που υπάρχουν στην Βοσνία Ζεγοβίνη. Τώρα, η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαλί για την εκπαίδευση. Είναι περίπλοκο ε, και πολιτάρχο το πλαίσιο και το Φεβρουάριο του 2003 ξεκινήσαμε δράσεις με, σε δύο άξονες με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Η πρώτη δράση είναι η κατάρτιση και εκπαίδευση των στρατιωτικών του Μαλή και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει την, ε, την εκπαίδευση του πέμπτου τάγματος του στρατού του Μαλή 8 έχουμε προγραμματίσει, 3.000 στρατιωτικούς ε, έχουμε εκπαιδεύσει και Μάλιστα προσπαθούμε να κάνουμε τους στρατικούς του Μαλή να ε, ιδιοποιηθούν την επιχείρηση αυτή και να μπορέσουν να αναλάβουν στα χέρια τους το μέλλον τους. Και μάλιστα ελπίζουμε ότι θα εξασφαλίσουμε αυτή την εθνοτική πολυμορφία στο Μαλί και φροντίζουμε αυτό να το διαφυλάξουμε. Υπάρχει όμως και ένας άλλος πυλώνας της δράσης μας, γιατί οι αποστολές μας δεν είναι αμυγός αποστολές εκπαίδευσης, αλλά ε, αποστολές αρρωγής για την διαμόρφωση ενός νέου στρατιωτικού σώματος. Και αυτή, αυτό είναι το πρώτο τμήμα της αποστολής μας. Παρέχουμε συμβουλές στις αρχές του Μαλή που έχουν ζωτική σημασία και θα πρέπει να δούμε πώς οι αρχές του Μαλή κάνουν κτήμα τους και το στρατητικό και το πολιτικό σκέλος αυτών των συμβουλών που δίνουμε και είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο να οικειοποιηθούν αυτές τις αποστολές και για, μάλιστα πρόσφατα η αποστολή μας συμμετείχε σε ένα σεμινάριο του Υπουργείου Αμήνης του Μαλή με θέμα τη μεταμόρφωση, το μετασχηματισμό του στρατού. Συμβάλλουμε λοιπόν σε διάφορες πτυχές, την οργάνωση της διοίκησης, επιμελητία, συγκέντρωση πληροφοριών. Είναι πολλοί τομείς που τους επεξεργαζόμαστε μαζί και χάρη των ε, αρχών του Μαλή. Στη Σομαλία επίσης έχουν μια αποστολή εκπαίδευσης και παροχή συμβουλών. Ε, έχουμε ήδη αναπτύξει πλήρως την αποστολή μας στο Μογκαντήσιο. Μέχρι το τέλη του έτους 1.400 στρατιώτες ε, από τη Σομαλία θα έχουν εκπαιδευτεί στο στρατόπεδο Αλτζαζίρα, στο προάστιο του Μογκαντήσιο μετά τους 3.600 στρατιώτες που εκπαιδεύτηκαν στην Ουγκάντα από το 2010 μέχρι το 2013. Η εκπαίδευση των εθνικών ενόπλων δυνάμεων της Σομαλίας ε, αφορούν κυρίως τη διοίκηση, τη συγκέντρωση πληροφοριών, αλλά και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τα δικαιώματα του ανθρώπου και την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Ξεπερνούμε δηλαδή την ε, αμυγή εκπαίδευση μαχητών και όπως και στο Μαλί, στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός, η επανίδρυση ενός νέου στρατού που θα εξυπηρετεί και την κυβέρνηση αλλά και τον πληθυσμό της Ομαλίας και το Μαλί. Επίσης παρέχουμε στρατηγικές σύμβουλες στις αρχές του Μογκαντήσιο. Έχουμε στενή συνεργασία και με άλλους ε, φορείς που είναι παρόντες, ε, τα Ηνωμένα Έθνη, η Αφρικανική Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε, Ιταλία, η Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες που εμπλέκονται στη Σομαλία. Τώρα, δεν πρόκειται να κάνω απολογισμό διεξοδικό των διαφόρων αποστολών, αλλά θα ήθελα να πω ότι κατά τη γνώμη μας σε όλες τις ε, επιχειρήσεις είμαστε αποτελεσματικοί αλλά ταυτόχρονα και ευέλικτοι σε ένα πλαίσιο ασφάλειας που είναι ευμετάβλητο. Και σε, σε όλα αυτά τα θέατρα των επιχειρήσεων η αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαίων είναι ορατή και μάλιστα αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Απόδειξη, η απόφαση της Ισπανίας να πάρει τη σκητάλη από τη Γαλλία ε, και να ηγηθεί της ε, αποστολής εκπαίδευσης ε, στο Μαλί για τις επόμενες εβδομάδες. Και μάλιστα και άλλες χώρες μετά την Ισπανία θα διαδεχθούν στην ηγεσία αυτής της αποστολής. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η προθυμία και δείχνει ότι η αλληλεγγύη είναι μεγάλη και επίσης μεγάλη είναι η κατανόηση του ενδιαφέροντος αυτών των επιχειρήσεων και έτσι οι χώρες αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κινδύνων. Ένα άλλο στοιχείο του απολογισμού. Κατά τη γνώμη μου, η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας, η Ευρώπη της άμυνας, εκεί που δραστηριοποιείται, δεν δραστηριοποιείται παντού, έχει προστιθέμενη αξία, κάνει τη διαφορά και μάλιστα σε περίπλοκες καταστάσεις. Οι αρχικοί ΓΕΘΑ βέβαια έχουν ασχοληθεί και με άλλα θέματα για παράδειγμα σε εθνικό επίπεδο, σε διάφορους ε, συνασπισμούς, αλλά και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της ε, Διατλαντικής Συμμαχίας. Εγώ θα επικεντρωθώ στις προσπάθειες που κάνουμε στη Στρατητική Επιτροπή κατά τίμα των αρχηγών ΓΕΘΑ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τέσσερα σημεία. Το πρώτο είναι η αλληλεγγύη. Τη στιγμή που οι προπολογισμοί είναι αρκετά συρρυκνωμένοι, ιδιαίτερα οι, προπολογισμοί άμυνα, είναι δύσκολο για να μην πω αδύνατο για τα περισσότερα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν το στόχο του 2% του προϋπολογισμού για την άμυνα και 20% για τις επενδύσεις. Οπότε θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ε, μία φιλόδοξη αλληλεγγύη μεταξύ μας. Και αυτό θα είναι εποφελές για όλου μα και για τι 28 χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για το ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Δεν θέλουμε να έχουμε περισσότερε δαπάνε. Σίγουρα δεν θέλουμε να περικόψουμε τις δαπάνες, αλλά σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο ε, διαχείρισης αυτών των κονδυλίων. Όχι λοιπόν περισσότερες δαπάνες, αλλά καλύτερες δαπάνες και χρειαζόμαστε αποφασιστικότητα γι' αυτό. Αυτό είναι ε, το αντικείμενο του ε, εγγράφω πλαίσιο για τη συνεργασία στο σχεδιασμό της άμυνας. Ένα κοινό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, μεταξύ άλλων, γιατί εγκύπτει σε ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητο και μάλιστα βρίσκει σύμφωνος και τους αρχηγούς ΓΕΘΑ. Δεν θα πρέπει να ενδιαφερθούμε μόνο για τον εξοπλισμό κατά την άφηξή του, αλλά τι ικανότητες δημιουργεί αυτός ο εξοπλισμός και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του, της λειτουργίας του. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Έτσι θα εξασφαλίσουμε διαλειτουργικότητα στη χρήση μεταξύ των διαφόρων των σωμάτων του στρατού και όχι μια πολυμορφία η απόκληση που θα αποβεί βάρος μας στα διάφορα θέατρα των επιχειρήσεων. Γιατί αυτές οι αποκλήσεις στον εξοπλισμό μας δημιουργήσαν και προβλήματα και στο παρελθόν. Δεύτερον, θα πρέπει η κυριαρχία να φροντίσουμε να ασκείται εκεί που χρειάζεται, εκεί που απαιτείται και μόνο τότε. Πριν από 20 χρόνια είχαμε μια διοίκηση αερομεταφορών ε, η ιδέα μάλλον μιας διοίκησης αερομεταφορών μεταξύ πέντε χωρών θα ήταν αδιανόητη. Σήμερα όμως αυτή η ιδέα της βελτιστοποίησης και της αξιοποίησης των μέσων και της αξιοποίησης των μηχανισμών μας και των ε, εργαλείων μας, αλλά και η εκπόνηση μελλοντικών μοντέλων, αυτή η ιδέα γονιμοποιείται. Δεν θέλουμε βέβαια να τη μεγεθύνουμε υπερβολικά, να την κάνουμε υδροκέφαλη, αλλά θέλουμε να τροφοδοτήσει και άλλα φόρα. Και μάλιστα οι σκανδιναβικές χώρες αυτή τη στιγμή δημιουργούν μία δομή παρόμοια με αυτή της διοίκησης αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει οι χώρες μέλη να αντιληφθούν ότι οι συνεργασίες σε μικρές ομάδες, σε κλάστερ, είναι μια συνεργασία ευεργετική και μάλιστα δεν εμποδίζει τις χώρες αυτές να αντιληφθουν οτι οι συνεργασιε σε μικρες ομαδες σε κλαστερ ειναι μια συνεργασια ευεργετικη και μαλιστα δεν εμποδιζει τις χωρες αυτες να επικεντρωθουν στον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους, που στα θέματα των μεταφορών αφορά την συμβολή στην διαθέτηση κατεπηγουσών κρίσεων και φυσικά εκένωση των υπηκών, απομάκρυση των υπηκών από ε, ε, τα πεδία της κρίσης. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες και να έχουμε σύγκληση των ε, τρόπων ικανοποίηση των αναγκών. Δεν χρειάζεται να έχουμε ίδιους εξοπλισμούς, αλλά τουλάχιστον συμβατούς μεταξύ τους. Δεν μιλούμε εδώ για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού, αλλά θέλουμε τουλάχιστον ομοιόμορφα και ομοιογενή χρονοδιαγράμματα, ώστε ο τρόπος έκφρασης των αναγκών να είναι παρόμοιος. Οπότε αυτό το έγγραφο πλαίσιο για τη συνεργασία στον τομέα της, του σχεδιασμού της άμυνας έχει θεμελιώδη σημασία, γιατί αν εγκριθεί από τις πολιτικές αρχές μέχρι το τέλη του έτους θα δώσει ένα νέο δυναμισμό στη συνεργασία στα θέματα αμυντικού σχεδιασμού. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναλύσω είναι το έργο της Στρατιωτικής Επιτροπής σε στενή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Η Στρατιωτική Επιτροπή στηρίζει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Έχουμε συνεργασία σε πολλούς τομείς. Θα αναφερθώ σε δύο. Καταρχήν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας στηρίζοντας ε, τις επιχειρήσεις ε, μας δίνει μια ανεκτήμητη βοήθεια σε θέματα επιμελητίας, διοίκησης και ελέγχου κατά την έναρξη των επιχειρήσεων. Και χάρη στις συμφωνίες ε, που ισχύουν έχουμε πιο ελαστικό σύστημα δημοσίων προμηθειών και χάρη στην, στο μεγαλύτερο ανταγωνισμό που υπάρχει, μειώνουμε το κόστος. Συνεργαζόμαστε βέβαια με τον οργανισμό και για τις ε, ικανότητες ε, του μέλλοντος. Θέλουμε να αυξήσουμε την ε, διαλειτουργικότητα των στρατών μας στο μέλλον. Και μάλιστα αυτό το θέμα μας απασχολεί ιδιαίτερος και εργαζόμαστε άοκνα γι' αυτό. Και μάλιστα η Στρατιωτική Επιτροπή συμβάλλει ιδιαίτερα στο θέμα των μη επαδρομένων αεροσκαφών, των drones. Όπως είπα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα αέρια drones, γιατί εκεί έχουμε τις περισσότερες ικανότητες και μάλιστα χρησιμο... τις χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο. Και μάλιστα στη... στο Κονγκό και στο Βόρειο Μαλί τα Ηνωμένα Έθνη χρησιμοποιούν drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και επίσης και στην Ουκρανία χρησιμοποιούνται drones. Πέραν των πλατφορμών αναγνώρισης, των ε, δορυφόρων ε, παρατήρησης και των πολεμικών αεροσκαφών, τα drones αυτά έχουν αποδείξει τη σημασία του για θέματα μόνιμης επιτήρησης στα θέατρα επιχειρήσεων. Αρχίζουμε λοιπόν και τα χρησιμοποιούμε σε διάφορα θέατρα επιχειρήσεων. Έτσι, η Ιταλία χρησιμοποίησε κάποια drones ε, καταδιοκτικά για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες στην επιχείρηση UNAFOR στην Αταλάντα. Γι' αυτό και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας μας ζήτησε να της δώσουμε κάποιες προτάσεις ε, για χρήση στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα εργαλεία συγκέντρωσης πληροφοριών, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε και <coughs> ποιες είναι οι προτάσεις μας ε, για διάφορα πεδία επιχειρήσεων και πώς ε, θα αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε σε πραγματικό χρόνο και πώς θα τις ε, μεταδίδουμε. Άλλο σημαντικό θέμα, οι εταιρικέ σχέσεις. Προτεραιότητα στο έργο της Στρατιωτικής Επιτροπής, γιατί οι εταίροι μας έχουν υψηλές προσδοκίες, ιδιαίτερα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στη Γεωργία, για παράδειγμα, η Γεωργία μάλλον εξασφαλίζει την προστασία του, του αεροδρομίου του Μπαγκουή. Και είναι πραγματικά αξιόλογο το έργο τους και αξιέπαινο. Η Σερβία συνέβαλε σημαντικά στην παροχή ιατρικής περίθαλψης κατά τη μετακίνηση της αποστολής εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μογκαντήσιο στη Σομαλία. Οπότε θα πρέπει να εντάξουμε καλύτερα τους εταίρους μας στη στρατηγική μας για να αξιοποιήσουν και τις δικές μας εμπειρίες. Φυσικά θα πρέπει να καταλήξουμε σε δίκαιο επιμερισμό των ρόλων μεταξύ των μελών και των τρίτων χωρών. Και τέταρτο σημείο, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Για να ανταποκριθούμε στις πολυάριθμε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι δύο οργανισμοί, θα πρέπει να συνεχίσουμε την ενίσχυση της συνεργασίας μας. Από τη στιγμή της Σύλληψη των επιχειρήσεων και στη συνέχεια και να ενισχύσουμε την συνοχή μας σε ό,τι αφορά τις ικανότητές μας. Και μάλιστα η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Νιούπορτ ε, επενθύμησε την επιτακτική ανάγκη ε, για αισθητή πρόοδο. Έχουμε πολλές απειλές ανατολικά, νότια της Ευρώπης και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις υβριδικές προκλήσεις ε, μόνο με τον έναν ή τον άλλον οργανισμό, τον ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε συνεργασία μεταξύ τους και στη φάση της ανάλυσης αλλά και στη φάση του σχεδιασμού και της αντίδρασης. Ακατακλείδη ε, θα ήθελα να πω ότι από τη θέση σε ισχύ της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε ότι έχει γίνει παγκόσμιος παράγοντας ε, που μπορεί να επηρεάσει τα γεγονότα και να συμβάλλει στην διευθέτηση και διαχείριση των κρίσεων. Και οι αρχηγοί για ΕΘΑ χρειάζονται σήμερα ένα διαφωτισμό, ένα καλύτερο ορισμό των στρατηγικών προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το έγγραφο αυτό που θα καταρτιστεί μέχρι το 2015, όπως μας ζήτησε το Συμβούλιο του περασμένου Δεκεμβρίου, είναι πολύ σημαντικό. Και στα πλαίσια αυτό, αυτής της διεθνής κατάστασης ε, με πολλές αιστείες κρίσεων, το έγγραφο αυτό αποκτά όλο και ιδιαίτερη σημασία και θα είναι καταλήτης για νέες συνεργασίες, ενώ θα ε, διευκολύνει την έκφραση μιας νέας ελληνικής μεταξύ των Ευρωπαίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και καλό θα ήταν ε, να το μεταφέρετε κι εσείς ε, στους συμπολίτε σας. Γιατί η Ευρώπη είναι η στόφα από την οποία αποτελούνται τα Ηνωμένα Έθνη. Και υπάρχουμε μέσω της πολυμορφίας μας, αλλά και χάρη στην πολιτική βούληση των 28 κρατών μελών μας και άρα του συνόλου των Ευρωπαίων που εκπροσωπείτε κι εσείς, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Είναι πολύ μορφό το πλαίσιο στο οποίο ενεργοποιείται η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Και η διπλωματία είναι δυνατή μόνο όταν στηρίζεται σε μια στεναρή βούληση και μάλιστα σε κατάλληλου αμυντικού μηχανισμού που θα συμβάλλουν στο να επηρεάσουμε τα γεγονότα και να εξασφαλίσουμε την ειρήνη. Μπορεί να μακρηγόρησα λίγο, αλλά ήθελα οπωσδήποτε να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ιδέες που είχα. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε, στρατηγέ. Τώρα θα αρχίσει η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ, συντονιστή του ΕΛ και την Επιτροπή ΣΕΔΕ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Στρατηγέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Είπατε ότι οι απειλές συνδέονται άμεσα με την έκυρα ενό κράτου και βλέπουμε ότι αυτέ οι απειλέ είναι ολαιόνα και πιο φανερές. Ε, σίγουρα πιστεύω πως χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική ε, ε, διπλωματία, μια εργαλειοθήκη τρόπον Α η οποία θα αποτελείται και από πολιτικά μέσα και από στρατιωτικά μέσα για να καταφέρουμε να επιτύχουμε αυτό που επιθυμούμε γιατί όπως λέω πάντα ε, πρέπει να έχουμε όλο το φάσμα των ε, μέσων στη διάθεσή μας. Έχω ορισμένες παρατήρησεις και ορισμένες ερωτήσεις σε αυτά που είπατε. Καταρχάς, ε, μας είπατε ότι ο τομέας της άμυνας χρειάζεται περισσότερους πόρους. Και αν δεν καταφέρουμε να έχουμε αυτούς ε, τους ε, πόρους και κάποια κράτη-μέλη ήδη τους ε, διαθέτουν. Πρέπει τουλάχιστον να έχουμε μια, πολύ, μια πολιτική συμφωνία ανάμεσα στα κράτη για να μην περικοπεί περαιτέρω ο αμυντικός προϋπολογισμός. Γιατί αυτό σίγουρα δεν θα είναι κανένα καλό πολιτικό μήνυμα από πλευράς μας. Και δεν πρέπει να, το, να χρησιμοποιήσουμε τον αμυντικό τομέα για να κάνουμε αυτές τις ε, περικοπές που χρειάζονται. Τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά την, τον αμυντικό εξοπλισμό και τα σχέδια και τις ε, προετοιμασίες για την επόμενη ε, σύνοδο για τα αμυντικά ζητήματα το 2015. Μετά από τον σχεδιασμό για τον εξοπλισμό τι θα ακολουθήσει, πού θα εστιάσετε, ποια ε, θα ήταν κατά την άποψή σας μια αποτελεσματική διάθεση των ε, κονδυλίων στον αμυντικό τομέα. Επίσης ακούσαμε για τις διάφορες αποστολές ε, που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Εσείς έχετε την εντύπωση ότι ο υφιστάμινος μηχανισμός που έχουμε αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός Ατένα. Είναι αρκετός. Μπορούμε να πούμε ότι η σχέση κόστους και αποδοτικότητας είναι σωστή. Η εμπειρία μας, ε, μας δείχνει ότι χρειάζεται ριζικές αλλαγές αυτός ε, ο μηχανισμός. Τώρα όσον αφορά το Μαλί, έχω μία ερώτηση. Μας είπατε ότι πάνω από 3.000 στρατιώτες βρίσκονται εκεί και καταρτίζουν το, τους ε, του Μάλι. Χρειάζονται όμως σε κάποιες ε, συμβουλές, στρατηγικής και από ό,τι έχω ακούσει υπάρχει ανάγκη ε, παρέμβαση στο βόρειο τμήμα του Μάλι έτσι ώστε να βοηθήσουμε για να επικρατήσει η τάξη. Χρειάζεται λοιπόν κάποια στρατιωτική επέμβαση. Να υποθέσω δηλαδή ότι δεν έχει υπάρξει κάποια ε, στρατιωτική συμβουλή από μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος ε, αναφέρατε την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Στατιωτικής Αεροπορίας. Έχετε σκοπό να συμπεριλάβετε και αυτήν την υπηρεσία στις επιχειρήσεις σας. Είναι πολλές ερωτήσεις, αλλά ελπίζω να μου απαντήσετε σε κάποιες από αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ιωάνν Πάσκο από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω εδώ. Ξέρω πως αυτά που θα πω δεν είναι άμεση αρμοδιότητά σας, αλλά αφορούν περισσότερο πολιτικές αποφάσεις, τις οποίες εσείς φυσικά πρέπει να εφαρμόσετε. Θα κάνω όμως την ερώτηση όπως και να έχει. Εάν όλα πάνε τόσο καλά με τις επιχειρήσεις μας ε, με όλα τα project που έχουμε αναλάβει. Γιατί εμείς έχουμε δείξει τόση ανασφάλεια, τουλάχιστον στα ανατολικά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι όπως γνωρίζετε η κατάσταση εκεί δεν αντιμετωπίζεται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται πράγματα τα οποία στα οποία δεν έχει απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει λοιπόν ένα κενό. Και όπως είπα, φυσικά δεν είναι δική σας ε, η ευθύνη για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, αλλά των ε, πολιτικών αρχηγών. Και κάτι, ένα σχόλιο. Όταν μας είπατε ότι υπάρχει αυτή η απειλή διάχυτη την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Αυτά τα, τα έργα μπορούν να γίνουν πιο εύκολα αν συμμετέχουν πολλοί στην ε, διεξαγωγή τους. Για παράδειγμα, οι εναέριες ε, μεταφορές μπορούν όλοι να συμμετέχουν σε αυτές και να μοιραστούν τον ε, φόρτο εργασίας. Να υπάρχει δηλαδή μία κοινή στρατηγική. Όμως, όταν αυτή η απειλή αλλάζει μορφή και γίνεται διαφορετική. Το αν εγώ προσωπικά σαν κράτος θα συμμετέχω σε ένα project θα έχει να κάνει με το αν αυτό το project είναι μια απειλή έτσι όπως την έχω εγώ στο μυαλό μου. Αυτές λοιπόν τις ε, σκέψεις και τις αμφιβολίες ήθελα να μοιραστώ μαζί σας διότι διαχειρίζεστε πάρα πολλά project και θα πρέπει τουλάχιστον να έχετε την επίγνωση το ότι υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες και κάποιες ερωτήσεις και κάποια δυσταγμή για συμμετοχή από τα κρατημέλη. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πάσκου. Ο κύριος Τζέφρι Βανόρτερ από τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να συμπληρώσω κι εγώ σε αυτά που είπε ο Ιωάνν και να απαντήσω σε αυτό που είπες. Ένας από τους λόγους που αισθάνεσαι σε τόση ανασφάλεια είναι φυσικά για το ότι έχει... έχουμε χάσει την εστίαση. Το ΝΑΤΟ έχει χάσει την εστίασή του δεν έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την ε, αναζωγόνηση του ΝΑΤΟ, ανανέωση του ΝΑΤΟ και δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στις ε, κοινωνικές ε, δαπάνες, στην πρόνοια περισσότερο από ότι στην, στον τομέα της άμυνας και να περιμένουμε από τον φορολογούμενο να αναλάβει αυτόν τον τομέα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πιστεί η κοινή γνώμη για την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για μια ισχυρή ασφάλεια και για την ανάγκη των, που, ύπαρξη των ενόπλων δυνάμεων. Είναι κάτι που δύσκολα το καταλαβαίνουν οι πολίτες και πολλές φορές καταλαβαίνω το γιατί. Αυτή είναι η άμεση αντίδρασή μου σε αυτά που είπες, αλλά τώρα θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο στρατηγό. Όπως γνωρίζετε, πολλές φορές σε αυτήν την επιτροπή, από αυτά που έχουμε ακούσει, δεν νομίζω ότι ότι πρέπει να επιμένει η Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Επιτροπή. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Επιτροπή είναι μία απομίμηση του ΝΑΤΟ. Σε πολλά σημεία δεν συμφωνώ με το έργο της και πραγματικά πρέπει να πω ότι το επιτελείο σας πρέπει να βρει το χρόνο για να δει ποιες ευκαιρίες υπάρχουν για να δημιουργηθούν αποστολές και project τα οποία μπορεί να διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά που μας περιγράφεται είναι ακριβώς αυτά που κάνει το ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, μιλάτε για αμυντικό σχεδιασμό. Και όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, υπάρχει αμυντικό σχεδιασμός του ΝΑΤΟ από την ίδρυσή του. Όπως γνωρίζετε επίσης υπάρχει μια δέσμη δημιουργίας αμυντικών ικανοτήτων για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στα μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν το κάνει το ΝΑΤΟ. Γιατί επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρέπει να αρχίσει έναν συμπληρωματικό αμυντικό σχεδιασμό. Επίσης μας μιλήσατε για εταιρικέ σχέσεις και για συνεργασίες και υπάρχουν όμως τέτοιες συνεργασίες και στο ΝΑΤΟ από τότε που θυμάμαι. Βλέπω, για παράδειγμα, γαλλο... Ε, ε, στρατεύματα κοινά Γερμανίας και Βελγίου και κάτι πιο πρόσφατο, το πλαίσιο του ΝΑΤΟ για συνεργασία των εθνών στη δημιουργία διαφόρων ε, πακέτων αντιμετώπισης στον κόσμο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλουμε πραγματικά συμπληρωματική δράση από πλευρά της Ευρωπαϊκή Ένωσης, τότε πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε και να δούμε πραγματικά πού υπάρχει η προστιθέμενη αξία. Για παράδειγμα, ανθρωπιστική, ε, ανθρωπιστικές πτυχές, οι πτυχές ε, των ε, πολιτικών, πτυχές της διπλωματίας, της διαχείρισης ε, κρίσεων. Αυτή είναι οι τρόποι με τους οποίους, εάν ήθελε πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να βοηθήσει, παρά το να προσπαθεί να γίνει μια, μια στρατιωτική δύναμη, παγκόσμια στρατιωτική δύναμη. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, συνειδητοποιώ πως αυτές δεν είναι τόσο ερωτήσεις για εσάς, διότι εσείς ξέρω πως έχετε άλλη δουλειά να κάνετε και είμαι σίγουρο πώ την κάνετε πάρα πολύ καλά. Είναι μια ερώτηση για τους ε, πολιτικούς ε, ηθήνοντε. Προσπαθούμε δηλαδή να φτιάξουμε κάτι πολύτιμο με υλικά που δεν είναι πολύτιμα. Και κάτι που θα ήθελα τέλος να σας ε, ρωτήσω, το οποίο το ανέφεραν κάπως και οι συνάδελφοι. Αυτές οι αποστολές εκπαίδευσης που έχετε. Αν μας αναφέρατε το Μαλί, αλλά και η επιχείρηση στη Σομαλία, είναι επιχειρήσεις τις οποίες ε, κάνετε διάφορες ε, ενημερώσεις, ε, εκπαιδεύσεις, επαγρύπνησης και είμαι σίγουρος πως έχουν κάποια χρήση, ωστόσο δεν είμαι σίγουρος ακριβώς σε ποια χρήση. Αυτές οι εκπαιδευτικές επιχειρήσεις δεν είχαν την επιτυχία που έπρεπε. Και βλέπουμε ότι, όπως και στη Σομαλία, αλλά και στο Μάλι, αυτές οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή διαλύονται. Και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια είναι τα συμπεράσματα που εσείς εξάγετε για την αποδοτικότητα αυτών των εκπαιδευτικών αποστολών. Ξέρω ότι θέλει να απαντήσει ο κ. Πασκού. Θα συμφωνήσατε να μιλήσετε μετά τους συντονιστές. Μικρός γύρος είναι. Και θα ήταν φρόνιμο. Δεν θα ήθελα να έχουμε μια, ένα μακρύ διάλογο. Και κρατάτε και την, ε, το αίσθημα ευτυχίας του υποστρατήγου έχουμε υποχρεώσεις και έναντι των ε, εταίρων μας της Ανατολικής Ευρώπης. Κυρία Μποντήλ Καμπάγιας, παρακαλώ. Στα Σουηδικά να μιλήσω. Έχω μία ερώτηση για την ε, από κοινού χρησιμοποίηση των πόρων. Το pooling and sharing. Πήραμε 300 τέτοιες προτάσεις, αλλά από ό,τι κατάλαβα υλοποιούνται 10-12. Πώς προχωρά η διαδικασία αυτή. Και κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για την κεντροαφρικανική δημοκρατία, το Μαλί και την Σομαλία. Όταν παρεμβαίνουμε σε μια στρατιωτική σύραξη με, στρατιωτικούς, ε, με στρατιωτικά μέσα ή τα άλλα πέτυχαν, στέλνουμε στρατιωτικές δυνάμεις. Το καθήκον μας ωστόσο είναι να δημιουργήσουμε και μια βιώσιμη ειρήνη χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω στρατιωτικέ δυνάμεις. Αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος μας. Καταλαβαίνω ότι η Ένωση το έχει και αυτό ως στόχο. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω συγκεκριμένα τι δουλειά κάνετε, τι έργο κάνετε στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στο Μαλί τι κάνετε για να αυξηθεί, να αυξηθούν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που χρειάζεται η χώρα αυτή για να μπορέσουμε να λύσουμε τους, να διαλύσουμε τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η σύγκρουση. Με άλλα λόγια, τι κάνετε για να, για να μην χρειαστείτε να μείνετε και να μην επανέλθετε. Σομαλία τώρα και το Αταλάντα. Από ό,τι κατάλαβα, εποπτεύεται και τα αλλιευτικά σκάφη. Πώς γίνεται αυτό πρακτικά, ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι εκεί γίνεται και πολύ μεγάλη παράνομη αλία. Ευχαριστώ κύριε Λόιζινγκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρήσετε τους κανόνες αυτής ε, της αίθουσας. Με ακούτε. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να τηρείτε τους κανόνες αυτής εδώ της αίθουσας όσον αφορά την δική μου πολιτική ομάδα και στο παρελθόν πάρα πολλές φορές Είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες ως πολιτική ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα και να σας ε, κάνω αυτή την παράκληση και επίσημα. Έχω δύο ερωτήσει και δύο τομείς. Καταρχάς όσον αφορά το, την Αταλάντα. Μας είπατε για αυτές ε, τις ε, θετικές επιπτώσεις που είχαν οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, στη... θα ήθελα να ρωτήσω πόσες επιθέσεις είχαν γίνει σε πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια πριν την επέμβαση της ε, Αταλάντα. Ε, επίτα όσον αφορά την πειρατεία βοήθησε η επιχείρηση Αταλάντα για να, ε, για να αλλάξει το πεδίο δράσης των πειρατών. Τώρα, Μα είπατε πως δεν υπάρχει ένας ενιαίο ευρωπαϊκός στρατός, αλλά πως τα κράτη-μέλη έχουν διαθέσει τις δικέ τους δυνάμει. Και είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να ξεχωρίσουμε τι ακριβώς θέλει το ΝΑΤΟ και τι ακριβώς θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις δυνάμεις. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι εκείνες που ζητούν να αυξηθεί ο αμυντικός προϋπολογισμός να ανέλθει στο 2% του ΑΕΠ. Στη Γερμανία ο μετικός προϋπολογισμός είναι στο 1,3% και αυτή η αύξηση θα είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ για να φτάσουμε το όριο του 2%. Βλέπετε εσείς να έχει δίκιο το ΝΑΤΟ σε, αυτές, σε αυτά τα αιτήματα. Επίσης να πω ότι σημαντικό για μένα είναι να υπάρχει διαφάνεια και όχι να πείσω τους ε, πολίτες να συμφωνήσουν σε αυτές τις αυξήσεις. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ. Μία απάντηση από τον Ιωάννη Πάσκο πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Έκπληξη είναι, δεν ήξερα ότι θα έπρεπε να απαντήσω, πάντως καλή έκπληξη. Ξεκινώ λέγοντας ότι το ερώτημά μου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι προτείνουμε μια αλλαγή φιλοσοφίας και συμμετοχής των μελών. Εγώ διατηρώ την φιλοσοφία μου, τη φιλοσοφία μου και μένω στην ομάδα μου. Αυτό που δεν να πω είναι ότι όπως ξέρετε η Ένωση έχει να κάνει με θέματα άμυνας. Το πρόβλημα ήταν ότι θα πρέπει με βάση τις νέες εξελίξεις να προσπαθήσουμε να κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας περισσότερο προς τις ανάγκες των χωρών, ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν ε, άμεσο κίνδυνο. Αυτή ήταν η ιδέα μου. Όταν, μπήκαμε, όταν μπαίνουμε στο ΝΑΤΟ, μπαίνουμε στο ΝΑΤΟ για να προστατεύσουμε την άμυνά μας απευθείας. Όταν μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπαίνουμε για πολλούς λόγους, αλλά μεταξύ αυτών και η ενίσχυση της άμυνας. Άρα η Ένωση έχει κάποια σχέση με την άμυνα. Υπάρχει περίοδος πριν τη σύγκρουση και περίοδος μετά τη σύγκρουση. Ε, περίοδοι κατά τις οποίες θα ήταν ενδεδειγμένη η δράση της Ένωσης. Πριν και μετά. Για τις χώρες που είναι ωστόσο χώρες της Ένωσης χωρίς να είναι μέλη του ΝΑΤΟ, θα ήταν σκόπιμο και τα θέματα της σύγκρουσης να αντιμετωπίζεται εδώ. Βεβαίως ξέρετε ότι το ΝΑΤΟ έχει ε, σκέψη να αναλάβει δράση σε άλλες χώρες, αλλά νομικά θα έπρεπε να έρθουν σε εμά για να, ζητήσουν, να συζητήσουν τα θέματα άμυνας. Το έχουμε συζητήσει επί νομίζω και δεν περιμένω ότι θα πείσω τον συνάδελφο κύριο Βανόντεν. Το έχουμε συζητήσει πρώτα από πο, πο, καιρό και νομίζω ότι θα θέλω να καταστήσω σαφές απλά τι ήθελα να πω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ στρατηγέ μου για την πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση που μας κάνατε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που ο Τζέφρι Βανόρντεν επέστρεψε με τις ίδιες πεπιθήσεις και τον ίδιο ίστρο. Είπε ο Τζέφρι ότι δεν πρόκειται ο Αμερικανός φορολογούμενος να αναλάβει όλες τις προσπάθειες για την Αμερικανική άμυνα. Ούτε φυσικά ο Ευρωπαίος ε, φορολογούμενος δεν θα τροφοδοτήσει την ε, αμερικανική αμυντική βιομηχανία. Γιατί όταν μιλάμε για την Ευρώπη, ε, ε, σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον ε, σημαντικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει μόνοι μας να υπονομεύουμε τη θέση μας για θέματα αμυντικής βιομηχανίας, γιατί αυτά τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Στρατηγέ μου, πολύ θα ήθελα να ε, συμμεριστώ την αισιοδοξία σας για την ανάλυση που κάνατε και πιστεύω ότι βρισκόμαστε ε, σε μια στιγμή όπου υπάρχει μια ένταση μεταξύ των μηχανισμών που διαθέτουμε και που έχουμε σε στρατιωτικό επίπεδο και σε αμυντικό επίπεδο και των σκοπών για τους οποίους θα έπρεπε να, να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα. Γιατί εδώ και 15 χρόνια έχουμε διάφορους μηχανισμούς και μέσα και βέβαια 15 χρόνια σε, υπό την ιστορική προοπτική είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να είμαστε επίοικείς. Έχουμε λοιπόν διάφορα μέσα για τη διαχείριση των κρίσεων, αλλά κυρίως είναι μέσα για διέξοδο από την κρίση και η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Μαλί για την εκπαίδευση είναι μια αποστολή που έρχεται παράλληλα μετά την κρίση και η επιχείρηση Αλτέα στη Βοσνία αφορά τα τελευταία στάδια της κρίσης. Πέραν της επιχείρησης Αταλάντα ίσως ε, και της ε, επιχείρησης ίσως στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία τα μέσα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας βοηθούν για το, την, το επίκεντρο της κρίσης. Τότε που δημιουργείται και η πιο φλέγουσα κατάσταση. Ενώ όλο και πιο κοντά μας έχουμε πραγματικούς πολέμους, πραγματικές συγκρούσεις, πραγματικές κρίσεις και άρα και οι απαντήσεις και οι αντιδράσεις μας θα πρέπει να είναι πραγματικές. Ουκρανία, Ιράκ, Σύρια, Λιβύη, σε λιγότερο βαθμό. Είναι όλες αυτές πραγματικές σειράξεις και συγκρούσεις και δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί δεν μας επιτρέπουν να αντιδράσουμε στρατιωτικά τουλάχιστον. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δράσουμε επί τούτου μετά τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Αυτό και υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των αποστολών μας που δεν είναι βέβαια περιτές, γιατί όντως ε, ε, έχουμε επαγγελματίες και ιδιαίτερα υπεύθυνου ε, ανθρώπους και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άχρηστες οι αποστολές μας και στη Σομαλία και στο Μαλή σίγουρα οι αποστολές είναι πολύ καλά οργανωμένες και το προσωπικό μας υψηλού επαγγελματισμού αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις γιατί το δόγμα το ίδιο το στρατηγικό μας περιορίζει. Για πολλές αποστολές έχω σοβαρές αμφιβολίες. Η αποστολή στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Ξέρετε ποια είναι η γνώμη μου για αυτή. Τη θεωρώ περίτη, άχρηστη. Το πρόβλημα στη Βοσνία Ριζεγοβίνη είναι κυρίως πολιτικό, διοργανικό, διεθνωτικό. Δεν έχει καμία σχέση με στρατιωτική διατήρηση της τάξης. Και η UNAFOR Αταλάντα, η εμβληματική ε, ε, αποστολή και επιχείρηση με πραγματική προστιθέμενη αξία, αλλά βρίσκεται σε ευθύνουσα πορεία και όλο και λιγότερες χώρες συμμετέχουν σε αυτή. Οι βασικές χώρες που τη στήριξαν αρχίζουν και απομακρύνονται σταδιακά, οπότε δεν μπορούμε για πολύ καιρό ακόμη να κρυβόμαστε πίσω από την Αταλάντα για να διατρανώνουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε στρατιωτικό επίπεδο. Τώρα κάποιες άλλες ε, δραστηριότητες εκπαίδευσης, αποστολές εκπαίδευσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλά οργανωμένες, αλλά τα αποτελέσματα θα τα δούμε μετά από μεγάλο διάστημα. Και είδαμε στο Μάλι τι έγινε πρόσφατα και προβληματίζομαι και εγώ με αυτά που είπε ο κύριος Γκάλερ. Και διαρωτώ με αν είναι σωστή, σωστός, σωστή στρατηγική ε, εφαρμογή όλων αυτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και τη μονομερή ανάμειξη μερικών ε, χωρών. Στην στρατιωτική, στη στρατιωτική επιτροπή στην οποία προεδρεύεται συζητήθηκε αυτό το θέμα, έγινε πρόταση για συλλογική απάντηση στα προβλήματα αυτά. Έγινε κάποια σχέδια για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, γιατί είναι φυσικά πολύ θετικό που μερικές χώρες ε, ε, παραδίδουν εξοπλισμό στο Ιρακινό Κουρδιστάν, αλλά υπάρχει σχεδιασμός για μια πιο συλλογική ευρωπαϊκή δράση στήριξης ε, προς τις κουρδικές δυνάμεις του Ιράκ. Αυτά, γιατί πραγματικά η κρίση είναι οξύτατη και νομίζω ότι θα πρέπει να δουν κάποιες ευρωπαϊκές απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Ντονζόν, κύριος Νάρτ. Ευχαριστώ. Ένα από τα στοιχεία του άρθρου 3 που προβλέπει τη σύσταση της Στρατηγικής Επιτροπής έχει θεμελιώδη σημασία. Στρατηγικό, στρατηγική πτυχή αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων. Εμένα με εκπλήσει η έκπληξη θα έλεγα. Για παράδειγμα έχουμε την έξαρση ε, του μουσουλμανικού, της μουσουλμανικής τρομοκρατίας ε, στο, ε, στο Μαλί και στο το ψευδοχαλιφάτο της οργάνωσης Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και τη Συρία. Έχετε μεγάλη στρατιωτική πείρα και ξέρετε στην κάτω από τη Σαχάρα Αφρική τι κατάσταση υπάρχει. Βέβαια, για 200 τζιπ χρειάζεται πολύ βενζίνη και στο Βόρειο Μαλί δεν υπάρχει καν βενζίνη. Χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα μεγάλα βιτιοφόρα για να εφοδιαστούν. Και στο Μαλί δεν υπάρχουν καν όπλα. Θα πρέπει να φτάσουν και έχουν φτάσει από τη Λιβύη. Ερωτώ λοιπόν, πώς είναι δυνατόν όταν ε, ανετράπει το καθεστώς του Καντάφη και γνωρίζοντας όλους τους στρατικούς εμπειρογνώμονες και εσείς ε, ως Γάλλος γνωρίζετε τι, έγινε την αντιπαράθεση Γαλλίας-Λιβύης ε, λόγω του Τσάτ. Ξέρετε ότι μεταξύ της Ματενσάρα στα Σοδανικά σύνορα μέχρι τον Γκάτ, το Μουρσούκ, ε, στην, στα Νίγερο-Λιβιανά σύνορα, πώς δεν έγινε μια ελάχιστη προσπάθεια από τις μυστικές υπηρεσίες για να αναχαιτιστεί η μεταφορά ε, βαρέων οχημάτων. Δεν μιλάω για το γιώτα της ερήμου. Μιλάμε για τεράστια φορτηγά που χρειάζονται. Τύπου Βελέρα ή Unimog. Δηλαδή ε, χρειάζονται προσιτές ε, διάβλοι. Και γνωρίζετε την κατάσταση στην υποσαχάρη Αφρική. Ξέρετε ότι αν κλείσουν τα περάσματα του Κοριστή και του Τομό δεν θα υπάρχει καμία πρόσβαση. Και στο νέο τη Αλγερία και στα σύνορα της Νιγηρίας ε, δεν είναι εύκολα να εντοπίσουμε κάποιες ε, εφοδιοπομπές. Εδώ μιλούμε για μαζική επίθεση, όχι για μεμονωμένες επιθέσεις. Οπότε στα πλαίσια του νέου ή ψευδοχαλιφάτου του Ιράκ μας εκπλήσει αυτή η του ιρακ μας εκπλησει αυτη η εκπληξη που νιώθουν οι δυτικοί για την ε, τεράστια στρατηγική και επιμελητιακή ικανότητα που έχει το, η οργάνωση Ισλαμικό κράτος. Έχουμε εκατοντάδες οχήματα, κάτι που προϋποθέτει τεράστια επιμελητιακή οργάνωση και αφοδιασμό σε βενζίνη, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβληση. Είναι αδύνατο να, να έπεσαν από τον ουρανό όλα αυτά. Έχω, τρέφω τεράστιο σεβασμό προς τους στρατιωτικούς, γιατί εσείς πληρώνετε με το αίμα και τον υδρότα σας επιτόπου τα πολιτικά σφάλματα. Δεν θέλω να επικρίνω την την, πολιτική, την στρατιωτική αποτελεσματικότητα. Τους πολιτικούς ε, έφομαι. Αλλά η πρόληψη θα πρέπει να είναι το βασικό παρέτο μιας στρατιωτικής, στρατιωτικής αποτελεσματικότητας. Πού βρίσκεται λοιπόν αυτή η στρατιωτική συγκέντρωση πληροφοριών, πώς ε, λειτουργούν οι στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες και μήπως πρέπει, αντί να πρέπει να καταστέλουμε και να αντιδρούμε, να επικεντρωθούμε στην πρόληψη χάρη σε καλύτερη οργάνωση των στρατηγικών μυστικών υπηρεσιών. Γιατί δεν μιλώ για ε, συγκεκριμένες και αποσπασματικές τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά για μαζικές και πολύ καλά οργανωμένες τρομοκρατικές επιθέσεις. Μακάρι να μπορούσα να είμαι πιο αισιόδοξο. Γνωρίζετε όμως κάλλιστα ότι αυτό που συνέβη στο Μαλί συνέβη χάρη στη λειτουργικότητα του, του γαλλικού στρατού και την παρουσία του στρατού του Τσάντ επιτόπου. Γιατί ο στρατός του Μαλή είναι αστείο, ε, ελάχιστης ή μηδενικής αποτελεσματικότητας και διαλύονται, σαν τη ζάχαρη μπροστά στον εχθρό οι στρατιώτες του Μαλή. Και στην περίπτωση της Σομαλίας ε, όχι απλώς ε, σαν τη ζάχαρη, αλλά περνάνε στις ε, φυλές τους όταν λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση αποτελεσματικών στρατιωτών και όχι ομοιόμορφων απλώς στρατιωτικών σωμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούκαν. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στατηγέ, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή για να μας δώσετε αυτές τις ε, πολύτιμες πληροφορίες για αυτά που κάνετε. Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, αρχίζουμε την ε, δεύτερη νομοθετική περίοδο μετά την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, όπου θεσπίστηκε και η θέση του είπα του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς πώς θα εκτιμούσατε τη συνεργασία σας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και υπάρχουν ε, διδάγματα που αντλήσατε από την συνεργασία σας ε, με την προηγούμενη και με την επόμενη είπατε εκπρόσωπο, την κυρία Μογκερίνη θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ η απάντησή σας, διότι σε μία από τις ομιλίες σας νωρίτερα, τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, μας αναφέρατε μία κάπως διαφορετική άποψη από αυτήν που αναφέρει ο κύριος Ντανζάν. Μας είπατε πως σας ανησυχεί η αποσύνδεση της ε, στρατιωτικής δράση από την Ευωσνία Ερζεγοβίνη και πως ε, θέλετε να πείσετε τα κρατημέλη να κρατήσουν μια στρατιωτική παρουσία εκεί. Ποια λοιπόν είναι η απάντησή σας ιδιαίτερα σε σχέση με τα σχόλια του κυρίου Νταντζάν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αγιάλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να θα πω ότι είναι η πρώτη συνάντηση στην οποία έρχομαι, έρχομαι από το χώρο των μεταφορών. Αλλά με ενδιαφέρει πολύ το θέμα που αφορά τις υποδομές τη στρατιωτική δράση που είχαμε πει ότι ιστορικά ήταν τα πιο αδύναμα στοιχεία σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση τη Ευρωπαϊκή Άμυνα. Θέλω την άποψή σα για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε νομοθετικά στην Ευρώπη ώστε να βελτιώσουμε και να προλάβουμε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την χρήση των, μη, των drones που θα έχουν μια εκθετική αύξηση από ό,τι φαίνεται λόγω του τρόπου χρησιμοποίησής τους και, και αν υπάρχουν ζητήματα ή θέματα όπου μπορούμε να παρέμβουμε προληπτικά. Δεύτερον, μια ερώτηση. Το θέμα εκπαίδευσης που αναφέρεται ε, στην περίπτωση του Μαρή, καταλαβαίνω και αυτά που είπε ο κύριος Νάτ, την αναμόρφωση, την ανα, δημιουργία στην ουσία ενός στρατού είναι κάτι που πρέπει να το δείτε ή όχι μόνο για το Μαλί αλλά γενικότερα όταν έχουμε δράσεις που χρειάζονται ανασύσταση ενός στρατού. Πώς ε, χρησιμοποιείτε εκ νέου την εμπειρία σας. Και μια τρίτη ερώτηση, το είπε ο κ. Ντανζάν. Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε προληπτικά εργαλεία. Είπε ο κύριος Ντανζόν ότι εμείς ε, δουλεύουμε κυρίως ε, σε αυτά που βλέπουμε, τουλάχιστον έτσι το βλέπουμε εμείς, σε θέματα μετά την κρίση, εκ των υστέρων. Η ερώτησή μου είναι, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να προλάβουμε χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία. Στο κείμενο πλαίσιο που ετοιμάζει η Επιτροπή σας ε, με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να μας δώσουν αυτή τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε δηλαδή μια δουλειά εκ των προτέρων νωρίτερα. Ευχαριστώ. Thank you. Marek Ο Marek Jurek. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον στρατηγό Ρουζιέ. Μας αναφέρετε πολλές στρατηγικές επιχειρήσεις που γίνονται στο όνομα υπό τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές, οι περισσότερες μάλλον βρίσκονται στην Αφρική. Στη Δυτική ε, κυρίως Αφρική, στη Σομαλία, στο κέρας της Αφρικής, ε, κατά πολέμηση της πειρατείας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και πραγματικά θα ήθελα να πατήσω φόρο τιμή στο έργο της Γαλλίας στη Δυτική Αφρική για την εξασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή αυτή γιατί η κατάσταση στην υποσαχάρη Αφρική είναι από τα πιο σημαντικά γεωπολιτικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Αναφέρατε μερικές φορές τον όρο αλληλεγγύη και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, γιατί πραγματικά η αλληλεγγύη είναι επιτακτική ανάγκη και θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις δράσεις μας. Ο κύριος Πάσκου είπε ότι θα περιμέναμε ίσως ε, ε, μεγαλύτερη, μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ανησυχία για αυτά που, από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για αυτά που συμβαίνει στα ανατολικά μας σύνορα. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε συγκεκριμένη στρατηγική. Και στόχος μας θα πρέπει να είναι ε, η λήψη υπόψη των αλλαγών που έγιναν μετά την ε, πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και αυτό χρειάζονται μια ένα στρατηγικό όραμα, γιατί δεν έληξε η επικράτεια της Ρωσίας απλώς με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί οι δομές υπάρχουν. Και μάλιστα έχουμε, έχουμε τα στρατητικά δόγματα της Ρωσίας της δεκαετίας του 1990 για, για τα σύνορά της και για την κυριαρχία των ε, λαών. Και επίσης ε, νωρίτερα στην ε, Στη δεκαετία του 50 είχαμε, μερικές, είχαμε πολλές διαφορές απόψεων και τώρα η Ρωσία παρεμβαίνει στα σύνορα και στα εσωτερικά γειτονικών χωρών υπό το πρόσχημα της ε, προστασίας ρωσόφωνων πληθυσμών. Ε, για παράδειγμα, θέλει να, να διαφυλάξει υποτίθεται κάποια μνημεία του Λένινε ή τη, τη ρωσική γλώσσα στην, ε, στην Ουκρανία. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να ενισχύσουμε τη δική μας ασφάλεια. Ε, φυσικά δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναλάβει ή να επικαλύπτει τις δράσεις του ΝΑΤΟ αλλά έχω κάποια αισιοδοξία και το θέμα της ε, συνεργασίας είναι σημαντικό, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι το θέμα της συμβίωσης και του επιμερισμού του έργου. Και η πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συμμετέχει και στο ΝΑΤΟ. Οπότε είναι εύκολο να έχουμε τη συμβίωση, τη συμβιωτική σχέση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, Βέβαια υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι ουδέτερες, αυτό θα πρέπει να το σεβαστούμε, αλλά νομίζω υπάρχει ε, έδαφος για τέτοια συμβιωτική σχέση. Είδαμε τι συνέβη πρόσφατα στη Γεωργία και μάλιστα προσπαθήσαμε να προτείνουμε την, ε, ε, την στρατηγική παρουσία της Ευρώπης σε κάποιες περιοχές που προσέρτησε η Ρωσία. Βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την διπλωματική ε, οδό που είναι πιο σημαντική, αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πω ότι η αλληλεγγύη δεν αποκλεί την ε, αποτροπή των απειλών. Βέβαια, ε, για την Πολωνία είναι πιο κοντά η Ουκρανία, ε, για τη Γαλλία είναι πιο κοντά η, κεντρική, η, η Αφρική. Υπάρχουν κάποιοι δεσμοί ιστορικοί και γεωπολιτικοί, αλλά φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση του εισβολέα και εδώ η θέση μας είναι, πρέπει να είναι ομόφωνη. Καμία από τις χώρες μας δεν θα πρέπει να εξοπλίζει τη Ρωσία με όπλα. Γιατί η Ρωσία έχει επιθετικές δράσεις ε, ή μπορεί να τις χρησιμοποιήσει κατά χώρο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι η Ρωσία συνέλαβε έναν ε, εστονό υπήκο στο έδαφος της Εστονίας υπό το πρόσχημα με την κατηγορία της ε, κατασκοπίας. Θα πρέπει να αναλάβουμε πιο ενεργό ρόλο. Έχουμε χάσει πολλές ευκαιρίες τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, κατά την ρωσική επέλαση στην Γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σαφχάουσεν. Έπειτα θα μιλήσω εγώ και μετά κλείνει ο κατάλογος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στρατηγέ, δύο θέματα συμφωνίας μας θέλω να αναφέρω. Πρώτον, υπάρχει όντως μια ευρωπαϊκή άμυνα η οποία δικαιολογείται διότι τα συμφέροντα και της Ευρώπης και της υπηρετικής ακόμα Ευρώπης δεν είναι προφανώς τα ίδια με αυτά της Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεύτερον, η δυναμική της ευρωπαϊκής άμυνας δικαιολογείται απόλυτα. Επίσης, υπογραμμίσετε ότι τούτο στηρίζεται στα κράτη και προφανώς εγώ συμφωνώ απόλυτα επ' αυτού. Το ερώτημα που σας θέτω είναι τα κράτη κατά την άποψή σας συμβάλλουν σήμερα επαρκώς στις αποστολές και τον επίγοντα χαρακτήρα τους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε επαρκή εργαλεία, επαρκή μέσα για, τους, για να τηρήσουμε τους στόχους άμυνας που έχουμε θέσει. Um, και εγώ και ο Μάρεκ Γιούρεκ είμαστε παιδιά της πολωνικής αλληλεγγύης, της Σολιντάρνος. Γι' αυτό και είμαστε πεπισμένοι για την ανάγκη επιβεβαίωσης της στρατηγικής επιλογής της υποστήριξης των χωρών που δίνουν μάχη για την ανεξαρτησία τους και για την εθνική τους κυριαρχία, που έδωσαν μάχη για την ανεξαρτησία τους και την κυριαρχία τους και θέλουν να τη διατηρήσουν μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Και θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε και να στηρίξουμε την επιλογή αυτών των χωρών. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία συγκεκριμένα θέματα. Χθες το απόγευμα γύρισα μετά από πολυήμερη επίσκεψη στο Κίεβο, όπου είχα συναντήσεις με πολλές προσωπικότητες και στην ουσία δεν είχαμε πρόσωπο της Ουκρανικής πολιτικής. Άσχετα με το αν πρόκειται για κυβερνητικούς κύκλους ή για κύκλους της αντιπολίτευσης. Όλοι οι ε, πολιτικοί εκπρόσωποι του Κιέβου και οι κυβερνώντε και της αντιπολίτευσης ε, ήταν ομόφωνοι υπέρ της ανάγκης στήριξης της Ουκρανίας και της ανεξαρτησίας της. Γιατί έγινε λόγος η επιθετική και μη επιθετική ε, και η ανάγκη τροφοδότηση αναζήτησης της Ουκρανίας με επιθετικά, με θανατηφόρα και μη θανατηφόρα όπλα και εξοπλισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Μάρεκ Γιούρεκ. Εδώ και πολλά χρόνια η συνεργασία στα πλαίσια της πολεμικής βιομηχανίας ε, υπήρχε μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μεταξύ μερικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας αλλά υπό το φως των εξελίξεων στην Ουκρανία. Και μετά την υπογραφή εκεχηρίας και κατάπαυση του πυρός από, τον, από την ρωσική επίθεση είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Θα ήθελα λοιπόν τα σχόλια του στρατηγού για τα θέματα αυτά. Επίσης, έχω μία ερώτηση για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη θεωρείτε ότι η συμφωνία του Dayton μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη για να δοθεί νέα πνοή στην πολιτική διαδικασία στη Βοσνία ριζεγοβινη και για να στηρίξουμε την ανάπτυξη της δημοκρατίας στη Βοσνία. Και τι γίνεται με, με το στρατό. Πού ανήκει ο στρατός. Και τρίτο θέμα, Συρία, Ιράκ και Ίσης, οργάνωση Ισλαμικό κράτος. Το απόγευμα θα έχουμε πολύ σημαντική συνάντηση, κοινή συνεδρίαση ΑΦΕΤ και ΣΕΝΤΕ για το θέμα αυτό, παρουσία του Ίσης σε Ιράκ και Συρία. Η οργάνωση αυτή Ισλαμικό κράτος είναι η πιο εύπορη τρομοκρατική οργάνωση του κόσμου. Και βλέποντας την ε, έκταση που έχουν λάβει οι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το γεγονός και να δούμε, να σταθμίσουμε τα μέσα που έχουμε, ο Δυτικός Κόσμος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αναχαιτήσουμε αυτή την εξέλιξη και την επέλαση και επέκταση του ίσης. Και φυσικά θα πρέπει να φροντίσουμε να αναχαιτιστεί αυτή η φυγή ε, νέων από την Ευρώπη στο και η στρατολόγησή τους στο Ιράκ και τη Συρία στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης. Στρατηγία έχετε το λόγο. Σα κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας που δείχνουν, αν και δεν χρειάζεται, ότι η επιτροπή σας είναι και πολύ σημαντική και ότι τα θέματα ενόπλων δυνάμεων και ασφάλειας πάντα ήταν σημαντικά, σήμερα είναι ακόμη περισσότερο. Να απαντήσω με τη σειρά των ερωτήσεων. Κύριε Γκάλερ, για τα τρία σημεία. Καταμερισμός του βάρους μεταξύ Ευρωπαίων είναι ένα μείζον θέμα και για τους αρχηγούς επιτελείων και για την επιχειρησιακή δομή. Στο ξεκίνημα, δεν να στο ξεκίνημα κάθε ιδέα παρέμβαση των ενόπλων δυναμών το πρώτο πράγμα ή ένα από τα πρώτα πράγματα που μπαίνουν στη συζήτηση είναι η έννοια, αυτό το θέμα της κοινή χρηματοδότησης, που βέβαια δεν λύνει τα πάντα, αλλά είναι ένας παράγοντας που επιτρέπει να βοηθήσουμε αφενός και να περάσουμε τη συζήτηση στα ουσιαστικά που δεν είναι χρηματοδότηση. Το πρόβλημα είναι ότι πολλά κράτη-μέλη που συμβάλλουν στις διάφορες αποστολές μας θέλουν να αλλάξουν κάπως την πορεία αυτή και στο πλαίσιο αυτό αυτό είναι που θα γίνει με την αναθεώρηση του, της συνένεσης Αθηνά που είναι υποσυζήτηση μεταξύ των κρατών μελών και που θα οδηγήσει μέχρι τέλους του έτους σε μια εξέλιξη περιορισμένη είμαι βέβαιος που ωστόσο θα επιτρέψει κάποια πόδια. Είναι παράλογο να έχουμε δυνάμεις που είναι εν αναμονή εμπλοκής τους, αλλά όταν και όταν ξεκινούν δεν είναι λογικό οι χώρες που στέλνουν τους στρατιώτες να έχουν και την απόλυτη πολιτική, οικονομική και ανθρώπινη επιβάρυνση. Η συζήτηση είναι ένα θέμα που δεν είναι μόνο δικό μας, γίνεται σε κάθε πολυεθνικό, σε κάθε πολυεθνική δομή. Είναι μια συζήτηση λοιπόν που προσπαθούμε να καλύψουμε σε όλες τις πλευρές της Βρυξέλλες. Μιλήσατε για το Μαλί. και την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας εκεί, ρωτώντας πώς συνοδεύουμε τους καταρτισμένους στρατιώτες μας στην άσκηση των αποστολών τους. Εμείς έχουμε δύο αποστολές κατάρτισης και στο Μαλή και στο που χρησιμοποιούμε την έννοια της προσέγγισης σε ένα έθνος, σε ένα κράτος πλαίσιο, γαλλική πρόταση, που σημαίνει ότι συνοδεύει τις ε, στρατιωτικές δομές που εκπαιδεύτηκαν στην ε, αρχή των δράσεών τους. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι οι δυνάμεις του Μαλή δεν, ε, δεν απέδωσαν στην ένοπλη σύγκρουση. Όχι, αυτοί που εκπαιδεύτηκαν από εμά απο, ε, λειτουργήσαν αποτελεσματικά και όπως έπρεπε. Η προβληματική της εμπλοκής είχε να κάνει με την πολιτική στρατιωτική απόφαση του τι πρέπει να γίνει πού αφενός και δεύτερον την δομή, την ιεραρχική δομή ε, λήψεως αποφάσεων που είχε προβλήματα στρατιωτικού χαρακτήρα. Αυτό είναι το κύριο ζητούμενο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί στην πλήρη αναδόμηση των ε, δυνάμεων του Μαλή. Οι δύο παράμετροι που αναφέρεται, κατάρτιση στρατιωτών και συμπεριφορά, συμπεριφορά ατόμων και συλλογική συμπεριφορά με επίγνωση ότι κάθε δράση τους έχει άμεση επίπτωση στο έθνος, την κυβέρνηση και τους συμπολίτε τους. Η συμπεριφορά λοιπόν, η ατομική συμπεριφορά σε ένα συλλογικό πλαίσιο των καταρτισμένων αυτών στρατιωτών είναι απόλυτα ικανοποιητική. Οι χώρες πολλές χώρες που μετέχουν στην αποστολή στο Μαλή δεν πρέπει να ντρέπονται για την κατάρτιση που ε, παρέχουν. Στο επίπεδο συμβουλίου είμαστε, στο επίπεδο συμβουλευτικής είμαστε ακόμα σε αρχική φάση, ίσως σε μεταγενέστερο χρόνο, είναι ένα μεγάλο ζήτημα, πρέπει πρώτα να προχωρήσουμε στις πρώτες, στα πρώτα στάδια. Μην ξεχνάτε ότι στον βορρά του Μαλή εμπλέκονται πολύ και τα Ηνωμένα Έθνη που με μια σειρά ε, στρατιωτικών ε, δομών ε, ασκούν και δραστηριοποιούνται στην ανικοδόμηση και την αποκατάσταση της τάξης με, σε στενή συνεργασία και με μας. Σομαλία. Σε ό,τι αφορά την συνοδεία των στρατιωτών, η αποστολή κάνει την συνοδευτή αυτή. Οι στρατιώτες που ε, κατατίζουμε έχουμε κατατήσει και είναι σε ένας όπου συνεχίζουμε να κάνουμε πρόοδο για να μπορέσουμε να δούμε την υλοποίηση των δράσεων που κάνουμε. Είναι ένα περίπλοκο θέμα στη Σομαλία όπως γνωρίζετε. Αερομεταφορές. Λίγα κράτη της Ένωσης εμπλέκονται σε αυτό και είναι λογικό. Το, το απαντώ στον κύριο Πασκού. Είναι λογικό διότι δεν μπορεί να γίνουν περισσότερα στις αερομεταφορές. Sky Team, Star Alliance, αυτό ισχύει παντού. Το Sky Team, Star Alliance δεν μπορεί να έχει όλες τις εταιρείε. Το ίδιο ισχύει και με εμά. Ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι κάθε κυβέρνηση, αν χρειαστεί, θα μπορεί να ξέρει ότι θα έχει ε, διαθέσιμα ε, αεροσκάφη. Εμείς έχουμε πέντε χώρες, αλλά η Γαλλία μπόρεσε να κάνει τις δράσεις, στη οποία μετέχει στην ομάδα αυτή, μπορεί να κάνει τις δράσεις της στο, στη Λιβύη, το Μαλί, δηλαδή ο καταμερισμός του βάρους, που έχει να κάνει με την κίνηση προσωπικού, τη μεταφορά των, ε, της επιμελητίας είναι δουλειά και των τεσσάρων άλλων κρατών μελών. Η ελεγγύη λοιπόν εκφράζεται μέσω αυτού του τρόπου πολύ συγκεκριμένα. Κύριε Πασκού, ως προς την ερώτησή σας για το τι μπορεί να κάνει η ΕΠΑ για να καθησυχάσει τις χώρες που βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη. Προφανώς η συνθήκη περιγράφει την στρατιωτική, ε, τον στρατιωτικό, να τους καθησυχάσει στρατιωτικά. 28 χώρες της Ένωσης έχουν δεσμευτεί σε αυτό, είναι στη συνθήκη. Υπάρχει ένας τομέας ωστόσο που πρέπει να προχωρήσουμε, είναι η ρήτρα λεγγύης. Το λέω αυτό διότι η ρήτρα αλληλεγγύη συνδέεται ή τεσπον λοιπόν συνδέεται από πολλού αποκλειστικά μόνο σε θέματα θεομηνιών. Οι ασύμετρες απειλές που αντιμετωπίζουμε, η, η αυξανόμενη ανάδειξη των προβλημάτων στις κυβερνοεπιθέσεις και άρα οι ανάγκες κυβερνοάμυνας οδηγεί στο να σας πω ότι η χρήση μη στρατιωτικών όπλων για αποσταθεροποίηση μιας ευρωπαϊκής χώρας ενισχύονται. Και σε τέτοιες δραστηριότητες δεν μπορεί να κάνει κάτι η Ατλαντική ε, Συμμαχία διότι είναι μια μη στρατιωτική παρέμβαση κατά βάση στην οποία μπορούμε να συμβάλλουμε οι στρατιωτικοί. Επίγει λοιπόν να αναρωτηθούμε για τον τρόπο που θα επέτρεπε αν χρειαστεί μια μέρα που ελπίζω ποτέ να μην γίνει να έχουμε μια έκφραση ευρωπαϊκής ελεγγύης σε ένα πλαίσιο ασύμετρων μη στρατιωτικών απειλών, απειλών που πιστεύω ότι υφίστανται. Κύριε Βαν πάντα χρήσιμο να επικοινωνούμε και να βλέπουμε και να ακούω αυτά που λέτε, αλλά να σας πω κάτι. Γιατί τη συζήτηση δεν υπάρχει ανταγωνισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Όταν βλέπω τους ε, επικεφαλείς των, των ενόπλων δυνάμεων, των στρατιωτικούς, φορούν την εθνική στολή τους. Δεν, δεν γνωρίζω ούτε έναν Γάλλο, Βρετανό, Ισπανό ε, στρατιωτικό που να έχει σήμα ΕΕ. Της χώρας του το σήμα έχει, τα, οι χώρες τους τους εμπλέκουν στην α ή β δράση γιατί το θέλουν, είναι σκόπιμο ή πρέπει. Ποτέ το ΝΑΤΟ δεν εξέφρασε βούληση να πάει στο Μαλί ή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ούτε έχει τα εργαλεία να κάνει αυτά που κάνει η στην κεντροφρικανικη δημοκρατια ουτε εχει τα εργαλεια να κανει αυτα που κανει η αταλαντη ούτως ή άλλως ε, η Αταλάντη δείχνει, είναι, είναι η συνέχεια μιας δράσης στα ε, στην χερσαία Σομαλία, μια ε, δράση που δεν είναι μόνο δράση στρατιωτική αλλά που προσπαθεί να ενσωματώσει τους ε, πειρατές. Στον έμπολα έχουμε κάνει πολύ καλή δράση για να ευαισθητοποιηθούν όλοι εμπλεκόμενοι ζητώντας ε, και τονίζοντας την ε, ανάπτυξη των προβλημάτων, ε, την ανάπτυξη των δράσεων για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής, γιατί μας έστειλαν τα στοιχεία ή οι υπεύθυνοι, οι ιατρικοί υπεύθυνοι του στρατού. Η οι υπευθυνοι οι ιατρικοι διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως φτιάχνεται είναι πολύ χρήσιμη η ΕΠΑΕ κάνει αυτά που είναι σύνθετα. Εμείς οι στρατιωτικοί όταν δουλεύουμε στο πλαίσιο της ΕΠΑ δεν είναι κάτι απλό για μας, διότι είμαστε ένας δρόν μεταξύ άλλων. Το ξέρουμε, το σεβόμαστε και το ακολουθούμε. Αυτό είναι και το, το θετικό στοιχείο μας. Κύριε Καβανάν, για το pooling and sharing, τη συγκέντρωση και κοινή διαχείριση των πόρων. Ένα από τα προβλήματα του pooling and sharing είναι το ότι ότι πηγαίνουμε προς το άγνωστο, βαδίζουμε προς το άγνωστο και είναι δύσκολο να πείσουμε τις πολιτικές αρχές και κυρίως τα Υπουργεία Άμυνας ή τα Υπουργεία Εξωτερικών ή τους αρχηγούς ΓΕΘΑ ότι έχει νόημα αυτή η συγκέντρωση και η κοινή αξιοποίηση των ε, πόρων. Γι' αυτό και αρχικά είχαμε έναν ατέρμονο κατάλογο ε, που ήταν σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά τελικά καλύτερο είναι να συγκεντρωθούμε σε συγκεκριμένα θέματα, σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Πάντως ε, και στο ΝΑΤΟ έχουμε pooling and sharing και smart defense και εκεί πραγματικά έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο. on ερώτηση για το Ιράκ και τη Συρία. Ρωτήσατε κύριε Ντανζόν τι κάνουμε εκεί. Η Στρατιωτική Επιτροπή προσπαθεί να αφυπνίσει τους πάντες για να συνειδητοποιήσουν τις προκλήσεις και τα διακυβεύματα. Η γνώση και η εκτίμηση της ε, κρίσιμης κατάστασης ε, δεν είναι κοινή παντού. Ο στόχος της Στρατιωτικής Επιτροπής είναι ε, να ενημερώνει τακτικά με πληροφορίες και να τροφοδοτεί τη συζήτηση στις πρωτεύουσε και στα Υπουργεία Άμυνας, ώστε αργότερα, όταν γίνει πολιτική συζήτηση, να αναλυθούν κάποιες δεσμεύσεις με εμπεριστατωμένη τη γνώμη που θα έχουν σχηματίσει. Κύριε Νάρτ, λέτε πού είναι οι στρατιωτικέ μυστικέ υπηρεσίε ε, και γιατί όλοι διαρριγνύουν τα ημάτια του για την έξαρση, για την επέκταση του ίσης. Υπάρχουν στρατιωτικέ μυστικέ υπηρεσίε. Το θέμα είναι πώ συμβάλλουν ε, τα κράτη-μέλη με την παροχή τέτοιων ε, πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών για να δούμε στη συνέχεια πώς θα εμπλακούμε. Και μια γενική ερώτηση για την πρόληψη. Πώς θα βελτιώσουμε την πρόληψη. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, προσπαθεί να διαμορφώσει ένα μηχανισμό για την ανάλυση της κατάστασης στις ε, εμπόλεμες περιοχές, ώστε να επικεντρωθούμε στην πρόληψη. Στηριζόμαστε στο έργο κάποιων think tanks, στο έργο των αντιπροσωπιών των 141 πρεσβειών και στην πραγματογνωμοσύνη όλων των επιμέρους φορέων, των μυστικών υπηρεσιών. Έτσι κάνουμε μια χαρτογράφηση του κόσμου για να εντοπίσουμε πού μπορούμε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες πρόληψης των κρίσεων είναι οι πρωτοβουλίε που αναλαμβάνονται και οι προσπάθειε που γίνονται. Η Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε κύριε Στρατηγέ για την παρουσία σα και για την ε, διεξοδική ανάλυση που μας κάνατε. Ολοκληρώσαμε αυτή τη συζήτηση, θα κάνουμε μια μονόλεπτη διακοπή και θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ με πολύ σημαντικούς καλεσμένους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 Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. allow me to... Κυρίε και κύριοι, επιτρέψτε μου να αρχίσω το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Μία παρουσίαση δηλαδή, η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με, την, με τα μέτρα διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εάν αυτό είναι ένας επαρκής μηχανισμός ανταπόκρισης στις υφιστάμενες προκλήσεις. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας σε αυτό το πάνελ. Ο κύριος Τίμο Κώστερ, διευθυντής στην Διεύθυνση Αμυντικής Πολιτικής και Εκανοτήτων του ΝΑΤΟ. Έπειτα ο κύριος Πέτρος Μαυρομιχάλης, από την αίθουσα επαγρύπνηση τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. και τέλος ο Τζο Κόλμοντ από το Ινστιτούτο Egmont για Διεθνείς Σχέσεις. Κύριε Κόσνα, έχετε το λόγο για να αρχίσετε την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ενημερώσω αυτήν την Επιτροπή για τις αποφάσεις που έχει λάβει το ΝΑΤΟ στην πρόσφατη σύνοδο του στην Ουαλία σχετικά με την συλλογική άμυνα και όχι μόνο. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι ενώπιον σας σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την ε, δημιουργία στήριξη από το κοινό. Για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό, χρειάζεται ένα ειλικρινής και συνεχής διάλογο ανάμεσα στους διάφορους φορείς. Υπάρχουν πολλές σημαντικές αποφάσεις ε, που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ασφάλεια που ελήφθησαν στη Σύνοδο στην Ουαλία. Θα συνεχίσουμε Λοιπόν, ως ΝΑΤΟ να θεωρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση έναν σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό εταίρο. Αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν οι ρόλοι και αυτή τη στιγμή το, το τοπίο της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει και αυτό. Το ΝΑΤΟ λοιπόν έχει δείξει την δυνατότητά του και την πρόθεσή του να ταποκριθεί στην αυτή πραγματικότητα και να διασφαλίσει ότι η Βεροεκλαντική Συμμαχία θα παραμείνει έτοιμη και ικανή να αμυνθεί οποιασδήποτε απειλή. Σήμερα το πρωί θα επικεντρωθώ στο, στο RAP, στο σχέδιο δράσης ετοιμότητας. Το σχέδιο δράσης αυτό του ΝΑΤΟ έχει δημιουργηθεί για να ανταποκριθεί ε, στις ε, απειλές που έχουν προκύψει από τη στάση της ε, Ρωσίας, την επιθετική στάση της Ρωσίας και τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία. Στόχος είναι να ανταποκριθεί σε όλες τις ε, προκλήσεις σχετικές με την ασφάλεια από όπου αυτές και αν προελθούν είτε από την Μέση Ανατολή, είτε από την ε, Βόρεια Αφρική, είτε από τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει υποστεί τον ΝΑΤΟ από το τέλος του ψυχρού πολέμου και στην ετοιμότητα και στην ικανότητα ανταπόκρισης σε οποιαδήποτε, σε οποιοδήποτε πολεμικό σενάριο. Στόχος είναι να στηρίξουμε τόσο τους συμμάχους μας όσο και τους υπόλοιπους εταίρους. Το σχέδιο αυτό έχει μέτρα αντιμετώπισης ε, όπως είπα, της προσαρμογής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στα νέα δεδομένα. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν γίνει. Πρώτα, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. Μία συνεχής παρουσία σε γη και θάλασσα στο ανατολικό, στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ, όπου θα συνεισφέρουν εκ περιτροπή όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Έχει στείλει το ΝΑΤΟ μέχρι στιγμή σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα το οποίο συνάδει απόλυτα με τις διεθνείς δεσμεύσει του. Τα μέτρα αυτά, τα διάφανα και ορατά μέτρα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ε, αμυντικούς. Είναι μέτρα ευέλικτα έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στι εξαφνικές αλλαγέ όσον αφορά το επίπεδο ασφαλεία. Τώρα, τα μέτρα προσαρμογή. Τα μέτρα προσαρμογή περιλαμβάνουν συστατικά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσει το ΝΑΤΟ για να αντιμετωπίσει τι προκλήσει στην ασφάλεια που μπορεί να ε, προκύψουν. Ε, μέτρα συλλογική ε, άμυνα και διαχείριση κρίσεων συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο δράση. Στόχος είναι η καλύτερη, καλύτερα ισορροπημένη αντίδραση του ΝΑΤΟ όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας και την ε, συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Γίνονται προσπάθειες για να γίνει εκ νέου αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας έτσι ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα ανταπόκρισης, να ενισχυθεί η δύναμη ανταπόκρισης του ΝΑΤΟ, να γίνουν βελτιώσεις στην ικανότητα να στηρίξει αέρια του συμμάχους του και να ενισχύσει τα μέτρα ελέγχου και διοίκησης. Θα ήθελα να σχολιάσω πολύ σύντομα τους ε, τομείς αυτούς, όσον αφορά την ικανότητα ανταπόκρισης. Αυτή η ικανότητα έχει αναπτυχθεί βασισμένη σε πολιτικές αποφάσεις και στρατιωτικές ικανότητες, ε, με στόχο την επέμβαση τη σωστή στιγμή στο σωστό μέρος, έτσι ώστε η αντιμετώπιση να είναι αποτελεσματική και αξιόπιστη. Για να ενισχυθεί λοιπόν η ικανότητα ανταπόκρισης, πρέπει να προσαρμοστεί στις αλλαγές του επίπεδου ασφαλείας. Αυτό προϋποθέτει τη λήψη της, ε, των κατάλληλων δράσεων, την δημιουργία της ε, δύναμης πολύ υψηλής ετοιμότητας ε, της TF, όπως λέγεται, η οποία δύναμη αυτή θα περιλαμβάνει πολλές χιλιάδες στρατεύματα εδάφους και θα μπορεί να αναπτυχθεί σε ε, διάστημα πολύ λίγων ημερών, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις εξαφνικές προκλήσεις που θα προκύψουν κυρίως στα ε, σύνορα του ΝΑΤΟ. Η δύναμη αυτή θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει πάρα πολύ γρήγορα και να ανταποκριθεί άμεσα έτσι ώστε να αναπτύξει μία αποτελεσματική δύναμη ελέγχου στα εδάφη των ανατολικών συμμάχων μας. Η δύναμη αυτή θα είναι παρούσα συνεχώς, θα έχει επανδρωθεί από τους συμμάχους ε, εκ περιτροπής. Επίσης, για να ενισχυθεί η άμεση δυνατότητα ανταπόκρισης και επέμβασης της ε, νέας δύναμης αυτής, θα χρειαστεί κατάλληλη υποδομή, κατάλληλος ε, αμυντικός εξοπλισμός ε, και τροφοδοσία και ένας σχεδιασμός μιας επίσης κατάλληλης στρατιωτικής βάσης. Η δημιουργία αυτής της νέας ομάδας θεωρήθηκε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα παρέχει μια εμφανή ένδειξη αλληλεγγύης και στήριξης. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης του ΝΑΤΟ, μέτρα ενίσχυσης του συμμάχους τους, ένα αέρια και μη έτσι ώστε να μπορούν να στηριχθούν οι σύμμαχοι, να μπορούν να αποτραπούν επιθέσεις των συμμάχων και να μπορούν οι σύμμαχοι να αμυνθούν κατάλληλα. Επίσης, προβλέπεται η ενίσχυση της ναυτικής δύναμης του ΝΑΤΟ στα πλαίσια της ε, εφαρμογή ε, της ε, αμυντικής στρατηγικής. Στα μέτρα λοιπόν αυτά θα υπάρχει μία μόνιμη ναυτική δύναμη η οποία θα στηρίζει όχι μόνο τους συμμάχους αλλά και τα μέτρα επαγρύπνησης όσον αφορά την στρατιωτική ετοιμότητα στη θάλασσα και επίσης θα υπάρχουν και συμπληρωματικές δράσεις της δύναμης αυτής στην Ευρωπαϊκή θαλάσσια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενισχύσεις αυτές ε, τι απαιτούν. Απαιτούν συγκεκριμένα επιχειρησιακά ε, σχέδια τα οποία θα απαιτούν με τη σειρά τους ε, κατάλληλες δυνάμεις που θα τοποθετηθούν σε στρατηγικά στιγμή στην επικράτεια του ΝΑΤΟ και θα είναι έτοιμα να αναλάβουν δράση. Για να γίνει αυτό, αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε και αναπτύσσουμε ένα μόνιμο σχέδιο άμυνας, το οποίο είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής μας. Τέλος, οι ενισχύσεις χρειάζουν, χρειάζονται επίσης κατάλληλο σύστημα πληροφοριών και ανταπόκρισης αρκετά ευέλικτο έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα τα ενδεχόμενα καθώς επίσης και ένα σύστημα ε, και ελέγχου. Πού βρισκόμαστε τώρα ως προς την εφαρμογή όλων των σχεδίων αυτών. Πού βρισκόμαστε λοιπόν όσον αφορά την υλοποίησή τους. Τα μέτρα αυτά του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε ισχύ εδώ και αρκετό καιρό και θεωρούνται πλέον βασικά συστατικά στοιχεία της στρατηγικής του ΝΑΤΟ τόσο σε εύρος όσο και σε διάσταση. Υπάρχουν και κάποια συμπληρωματικά μέτρα επίσης. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν διαθέσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε μια ε, πρωτοβουλία συνεργασία με, τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Όλα αυτά τα μέτρα συνοδεύονται και από ε, μελέτες για τα νέα είδη πολέμου, όπως για παράδειγμα τον υβριδικό πόλεμο και τα πιο επανδρομένα σκάφη. Επίσης το σχέδιο αυτό παρέχει τα κατάλληλα μέσα στους ε, συμμάχους έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε αλλαγές του επίπεδου ασφαλείας στην επικράτεια της ε, συμμαχία. Ευχαριστούμε κύριε Κωστέρ. Τώρα ο κύριος Πέτρος Παυρομιχάλης που είναι προϊστάμενος τμήματος <clears throat> της αίθουσας επαγρύπνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος ε, για να μας ενημερώσει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πιθανά τη σχέδια για να ενισχύσουμε αυτά τα μέτρα εδαφικής διαβεβαίωσης. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ο ρόλος μου ως προϊστάμενος τμήματος της αίθουσας επαγρύπνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάπως περιορισμένο. Το τμήμα μου, η υπηρεσία μου, είναι το σημείο επαφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από μια σημαντική καινοτομία της συνθήκης της Λισαβόνας, δηλαδή την εισαγωγή της ρήτρα αλληλεγγύης. Και αυτή θα σας παρουσιάσω σήμερα. Η ρήτρα αλληλεγγύης συνιστά μια σημαντική καινοτομία της ε, τελευταίας αναθεώρησης ε, της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύπτεται στο άρθρο 222 και προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δρουν από κοινό υποπνεύμα αλληλεγγύης αν ένα κράτος μέλος ε, βρεθεί στο στόχαστρο μιας τρομοκρατική επίθεση ή ε, επλήγει από μια θεομηνία ή ανθρωπογενή καταστροφή. Στην τρίτη παράγραφο, το άρθρο αυτό προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος θα πρέπει να καταθέσουν κοινή πρόταση ε, να την υποβάλουν στο Συμβούλιο, το οποίο θα, θα αποφασίσει πώς θα εφαρμοστεί η ρήτρα αλληλεγγύης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έγινε ήδη και μετά από ε, μήνες συζητήσεων το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέτει στις 24 Ιουνίου του 2014 μία απόφαση για τις διατάξεις εφαρμογής προκειμένου να εφαρμοστεί η ρήτρα αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βασικά στοιχεία του μηχανισμού που ενέκρινε το Συμβούλιο είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, η επίκληση της ρήτρας αλληλεγγύης αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του θυγόμενου κράτου μέλους, δηλαδή του κράτους μέλους που έχει πληγεί είτε από τρομοκρατική επίθεση είτε από θεομενή ανθρωπογενή καταστροφή. Με βάση τους μηχανισμούς και τις χείουσε διαρθρώσεις ε, προβλέπεται στενή συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων και των κρατών μελών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων που θα πρέπει από κοινού να παράσχουν μια άμεση, συνεκτική και αποτελεσματική αντίδραση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς και τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και η ΠΑΤΗ εκπρόσωπος, με τη βοήθεια της ΑΕΔ θα εντοπίσουν όλους τους ενωσιακούς μηχανισμούς και μέσα και ικανότητες που μπορούν να να συμβάλλουν καλύτερα στην αντιμετώπιση της κρίσης και καλούνται να αναλάβουν όλα τα μέτρα που τους επιτρέπει η αρμοδιότητά τους. Επίσης, ε, ενεργοποιείται άμεσα και η διάταξη για την IPCR, για την, για την αντίδραση σε κρίση, που υιοθετήθηκε επίσης τον Ιούνιο του 2014 το Συμβούλιο και έτσι επιτρέπεται η ανάμειξη, η εμπλοκή των πολιτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η στρατηγική, ε, ο στρατηγικός προσανατολισμός της δράσης προς όφελος των ε, ε, πληγέντων κρατών μελών. Με την επίκληση της Ρήτρας αλληλεγγύης, το Κέντρο Συντονισμού για Αντίδραση στην Κρίση, που διαχειρίζεται η Γενική Διάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έχει επαφές με τα σημεία τα γραφεία επαφή των κρατών μελών 7 ε, μέρες, 24 ώρες 24 ώρα 7 μέρες τη εβδομάδα και θα έχει επαφή με όλα τα δίκτυα της Γενικής Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης Home και, Home και σάνκο καθώς και με, το γραφείο, με την αίθουσα επαγρύπνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης εν γέννη. Η ρήτρα αλληλεγγύης καλύπτει και εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις, ανάλογα με τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους. Και από αυτή την άποψη η ΕΙΕΔ έχει κάποιο ρόλο. Οπότε, όπου δει, η ύπατη εκπρόσωπος και οι υπηρεσίες της ΕΙΕΔ συμβάλλουν με την ανάληψη πρωτοβουλειών και την παροχή κατάλληλων πληροφοριών και στήριξη στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας αλληλεγγύης, η ύπατη εκπρόσωπος ε, κάνει ό,τι μπορεί για να εντοπίσει και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ε, για να αντιμετωπίσει καλύτερα την κρίση. Έτσι ε, θα πρέπει να εντοπίσει και ποιες στρατιωτικές ικανότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση κρίση με την υποστήριξη του στρατιωτικού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση θεομηνίας οι στρατιωτικοί πόροι μπορούν να συμβάλλουν και να στηρίξουν τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας ή τις μονάδες πολιτικής προστασίας. Η, είπατε εκπρόσωπος και υπηρεσίες της θα υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις επαγρύπνης και ανάλυσης κατάστασης προκειμένου να στηρίζουν το συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο στο Συμβούλιο. Η ε, θα πρέπει να είναι έτοιμη να παρέχει και πληροφορίες σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης και άλλες πληροφορίες με βάση την ανάλυση της κατάστασης μετά από πληροφορίες που λαμβάνονται από διάφορες πηγές ε, με κεντρικό συντονισμό από την αίθουσα επαγρύπνησης Ευρω... Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι εκπρόσωπος έχει και δικαίωμα πρωτοβουλίας. Μπορεί δηλαδή να υποβάλει προτάσεις και να ζητά ενεργοποίηση των στρατιωτικών ε, ικανοτήτων που θα υπερβαίνουν τις διατάξεις της ρήτρας αλληλεγγύης. Αυτό βέβαια θα ακολουθήσει τη νομική βάση και τις κανονικές συνήθειες διαδικασίες της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ο μηχανισμός της ρήτρας αλληλεγγύης δεν έχει αμυντικές επιπτώσεις. Δηλαδή δεν πρόκειται για μια αμυντική πολιτική για στρατιωτικό εργαλείο. Πρόκειται για μη στρατιωτικό εργαλείο, πολιτικό. Αν και σε μερικές κρίσεις όπως είναι οι θεομηνίες, χρησιμοποιείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο στρατός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η επιχείρηση είναι στρατιωτικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που μία αντιμετώπιση, η μία αντίδραση απαιτεί δράσει τη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτικης ασφαλειας η της ευρωπαικης πολιτικης ασφαλειας και αμυνας θα πρεπει να ληφθουν αποφασεις με βαση τι οικιε διαταξει τη συνθηκη για τετοιες διαδικασιες απαιτειται η ομοφωνη ληψη αποφασεων Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαυρομιχάλη. Ο κύριος Τζο Κόλμοντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πάντα είναι τιμή μου να με καλείτε εδώ, σε αυτό το κοινοβούλιο, σε αυτήν την επιτροπή, για να μιλήσω για ζητήματα ασφαλείας, αλλά και για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Άμυνας όσο και για τις σχέσεις μεταξύ της κοινή ε, αμυντικής πολιτικής και του ΝΑΤΟ. Ως ε, πολίτης αλλά και ως ε, στρατιωτικός εκτιμώ το έργο που κάνετε. Τώρα, ποια είναι τα διδάγματα που εμείς οι Ευρωπαίοι μπορούμε να αντλήσουμε από την, σύνοδο, την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να την, ε, να την θεωρήσω ένα μέρος ε, τριών ε, συνόδων. Την σύνοδο του Δεκεμβρίου σχετικά με την άμυνα και εκείνη που πρόκειται να γίνει μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της Συνόδου τη Ουαλία. Καταρχά η μερίσια διάταξη είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τα πρόσφατα γεγονότα, εάν όχι απόλυτα επηρεασμένη από αυτά. Και σίγουρα δεν ήταν γραφειοκρατική η διαδικασία κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε πέντε χαρακτηριστικά από την σύνοδο αυτή. Και θα επανέλθω σε αυτόν. Καταρχάς να πω ότι η Ρωσία δεν ήταν προσκεκλημένη. Ήταν δηλαδή πραγματικά προφανές, προφανής η απουσία της. Έπειτα, όχι μόνο στην αίθουσα, αλλά παντού υπήρχε και ένα άλλο φάντασμα που πλανιόταν εκτός από τη Ρωσία, ή το Ισλαμικό κράτος. Και περίπου το 60% της προσοχής των ε, προσκεκλημένων ήταν στην, στο Ισλαμικό κράτος. Τρίτον, η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε παρέμειναν προσκολλημένες στους στρατηγικούς τους στόχους. Και για τις Ηνωμένε Πολιτείε ο κύριος εταίρος, ο πρώτος τους εταίρος είναι η Ευρώπη. Οι στρατηγικές τους όμως προτεραιότητες βρίσκονται αλλού. Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και εκείνη παρούσα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα όμως είναι ποιοι ήταν οι στρατηγικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνοδο αυτή. Και πέμπτο και τελευταίο, στα πλαίσια της ε, συνόδου αυτής έλαβε χώρα ένας έντονος διάλογος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχε όμως να κάνει ούτε με στρατιωτική ζητήματα ούτε με το ΝΑΤΟ, αλλά με κυρώσεις και με αυτά που γίνονται στις Βρυξέλλες. Όλοι αυτοί οι λόγοι λοιπόν ε, απασχόλησαν πάρα πολύ τη σύνοδο στην ε, Ουαλία και προτού φτάσω στις συμπεράσματα θα ήθελα να αναπτύξω ορισμένους από αυτούς τους λόγους. Καταρχάς η Ρωσία και η κρίση στην Ουκρανία. Πράγματι, Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για την συλλογική άμυνα, για την υψηλή ετοιμότητα, αποτροπή και παροχή εγγυήσεων στον χώρο της άμυνας, ε, η προσοχή μας έχει στραφεί στη Ρωσία περισσότερο από ποτέ. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε έναν ψυχρό πόλεμο, διότι αυτή η ομάδα του ΝΑΤΟ είναι ικανή στον αριθμό. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε όμως ε, ήταν υπέρ αυτού του νέου συστήματος, διότι πιστεύουμε πως για τις Ηνωμένε Πολιτείε η παροχή εγγύσεων είναι αναγκαία, διότι δεν παρήχε μόνο εγγυήσεις και διασφάλιση στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και στους ε, εταίρους των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ασία. Επιπλέον, συζητήθηκε πάρα πολύ συλλογική άμυνα. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση της διαχείρισης κρίσεων, η οποία συζητήθηκε στην προηγούμενη σύνοδο. Έχουμε κατανοήσει πλέον ότι οι λεπτομέρειες της παρούσας κρίσης εντοπίζουν έναν οργανισμό, μία συμμαχία ή μία χώρα που πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Επίσης, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν την γενικότερη άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει γρήγορα αυτονομία. Και τέλος, αυτό που παρατηρώ εγώ είναι μια αυξανόμενη αντίληψη από όλα τα κρατημέλη πως πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα σοβαρά. Ωστόσο, δεν συζητήθηκε ένας οδικός χάρτης για μία αποτελεσματική συνεργασία ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ε, τομέα της, άμυτα, της άμυνας. Και αυτό πιστεύω πως πρέπει να είναι ένα από τα κεντρικά θέματα που θα απασχολήσουν τις ε, επόμενες συνόδους. Και τώρα συμπερασματικά θα ήθελα να πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη η μεγαλύτερη απειλή στην Ευρώπη δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτά που γίνονται εκτός της επικράτειάς τη. Πιστεύω πως η μεγαλύτερη απειλή είναι η αυξανόμενη αδυναμία εξαιτία του κατακαιρματισμού. Του κατακαιρματισμού στο εσωτερικό της Ένωσης. Υπάρχει καλή θέληση, αρκετή καλή θέληση. Υπάρχουν και πρωτοβουλίε. Και στο ΝΑΤΟ η λέξη που ακούγεται συνέχεια είναι η εφαρμογή. Εφαρμογή όλων αυτών ε, που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στην Ουαλία. Η εφαρμογή της έξυπνης άμυνας, του ε, πλαισίου για την αμυντική πολιτική. Και έχουν δημιουργηθεί αυτές οι ομάδες μάχης, όπως λέγεται, για να, το, να υλοποιήσουν αυτές τις αποφάσεις που περιέχουν πάρα πολλούς φορείς ε, και την αμυντική βιομηχανία. Είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και η συνθήκη της Λισαβόνας περιέχει πάρα πολλά πράγματα που χρειάζονται εφαρμογή και υλοποίηση. Ακούσαμε λίγο πιο πριν για την, ε, αμυντική, για την ρήτρα αλληλεγγύης. Υπάρχει όμως και στο άρθρο 44 ε, αναφορά στην αμυντική συνεργασία. Υπάρχει λοιπόν όλο αυτό το έργο που πρέπει να γίνει και υπάρχει και αυτή η καλή θέληση. Όμως, ε, αν κοιτάξουμε τα, τις ελλείψεις μας στον στρατιωτικό τομέα, θα δούμε ότι αυτό μας αποτρέπει από το να αποκτήσουμε αυτήν την ε, αμυντική αυτονομία στην Ευρώπη. Και δυστυχώς σε αυτόν τον τομέα δεν έχουν γίνει αρκετή πρόοδος. Και χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παρά να μοιράζεσαι την ανησυχία σου. Θα ολοκληρώσω λοιπόν λέγοντας ότι είναι αξιοσημείωτο ότι στο ανώτερο επίπεδο, σε επίπεδο αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων, ήταν ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνει στο ΝΑΤΟ, ότι πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αυτονομία που πρέπει να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν όμως αυτό μεταφράζεται σε έργα, τότε παρατηρούμε αυτόν τον ε, κατακαιρματισμό. Και ε, αυτό μπορεί να εξηγηθεί με έναν απλό τρόπο με το ότι λείπει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλεια στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αλλά τώρα πλέον γνωρίζουμε ακριβώς πώς ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές στην ασφάλεια. Όμως δεν γνωρίζουμε ποιος πρέπει να κάνει τι. Θα κλείσω λοιπόν λέγοντας ότι αυτή η στρατηγική ασφαλείας είναι αναπόσπαστη προϋπόθεση για να μπορέσουμε μαζί με τον ΝΑΤΟ να δημιουργήσουμε μια πραγματικά αποτελεσματική αμυντική στρατηγική. Τα κύρια λοιπόν στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση που εμποδίζουν αυτή τη δημιουργία είναι αυτές οι αδυναμίες. Αυτές οι αδυναμίες στην συνεργασία και στην αλληλεγγύη, τα οποία εμείς τα ίδια τα κράτη-μέλη έχουμε δημιουργήσει. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον, και εγώ, όπως και ο προηγούμενος στρατηγό, παραμένω αισιόδοξο. Αισιόδοξο διότι έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο εδώ και σύντομα θα έχουμε και μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πραγματικά ανυπομονώ να δω το έργο αυτού του κοινοβουλίου και το εμπιστεύομαι απόλυτα. Σας ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. Περνάμε στη συζήτηση. Θα ήθελα να σας παροτρύνω να υποβάλλετε ερωτήσεις στους καλεσμένους μας. Θα είναι πιο εύκολο και για εκείνους να απαντήσουν. Δεν κατάλαβα ποιος συντονιστής θέλει το λόγο. Ο κύριος Γκάλερ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε στο ίδιο τραπέζι ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε και την σύνοδο του Δεκεμβρίου, μετά το Δεκέμβριο είχαμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Αύγουστο. Είμαστε στο ημίχρον μεταξύ των δύο συνόδων κορυφής άμυνας της Ένωσης. Η ερώτησή μου είναι δεδομένων των εξελίξεων από την αρχή του χρόνου, ιδίω στην άμεση γειτονιά μας ανατολικά, αλλά και στις προκλήσεις στο Νότο, τι αξιολόγηση κάνετε ως ειδικοί και υπεύθυνοι για την κατάσταση. Θα παροτρύνουν την υλοποίηση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων που έχουν ε, τεθεί και στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι η εξανάγκης, η εξέλιξη, η δραματική εξέλιξη των γεγονότων που είδαμε θα οδηγήσουν σε πιο κοινή προσέγγιση ή σε μια κοινή ημερήσια διά, ε, διάταξη για να καλυφθούν τα ελλείμματα που υλοποιήσεις που διαπιστώσαμε. Ή υπάρχουν λίγα κονδύλια, υπάρχει απομάκρυση, τον είπα, υπάρχει διαφορία από πλευράς μας ε, λέγαμε στο παρελθόν. Αλλά τα άλλα δύο δεν υπήρχαν. Τώρα έχουμε και τα τρία. Και απειλές και απομάκρυνση των ΙΠΑ και οικονομικά προβλήματα. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν σήμερα εν ώψη και των επόμενων συνόδων κορυφής. Κύριος Πάσκου. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση προς τον κύριο Κώστα. Το, σα... το επίπεδο εξουσίας του ΣΑΚΕΡ συζητείται, είναι υποσυζήτηση, διότι κάποια πράγματα πρέπει να αποφασίζονται πολύ γρήγορα. Και αν έχουμε καταστάσεις όπου πρέπει να το εγκρίνουν όλοι, δεν είναι εύκολα πράγματα. Κατόπιν, δύο ερωτήσεις και ένα σχόλιο για τον κύριο Μαυρομιχάλη. Τι γίνεται με τις αμυντικές ανάγκες των μελών της Ένωσης που δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Είπατε, η αλληλεγγύη, η κρίτα αλληλεγγύης δεν καλύπτει στρατιωτικές καταστάσεις. Άρα αυτοί οι άνθρωποι ποιον θα πρέπει να... από ποιον πρέπει να ζητήσουν άμυνα. Μετά, Υπάρχει δυνατότητα να ερμηνευθεί, για παράδειγμα, η συνέπεια μιας επίθεσης σε μια χώρα ως ανθρωπογενής καταστροφή που θα ενεργοποιούσε τρίτα λεγγύς ή όχι. Ε, μάλλον όχι, καταλαβαίνω εγώ. Ήταν μια σαφής θέση ότι μη μπούμε σε αμυντικές παραμέτρους. Αυτό το σενάριο είναι εφικτό ή όχι. Ένα σχόλιο. Ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία λήψης απόφασης διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή καθιστάς, καθιστά άσχετη, μάταιη μια τέτοια κατάσταση. Μέχρι να υπάρξει ομοφωνία στο Συμβούλιο και το ένα και το άλλο μέχρι να φτάσουν οι ηγέτες στον ε, χώρο συζητήσεων, γιατί ξέρετε μπορεί έχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στις Βρυξέλλες. Πια σταυρό και αυτό Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να λάβει υπόψη και αυτές τις παραμέτρους. Ο κ. Βανόντεν, συντηρητική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. προς τον στρατηγό Κόλμαντς. Πάντα χαρά είναι να έρχεσαι εδώ πέρα να προσταθεί την είναι τα μη υπερασπίσιμα. Τώρα, στη Σύνοδο Άμυνας του Δεκεμβρίου. Ήταν μια απογοήτευση σε όσους είχαν ε, την ελπίδα μιας φιλόδοξης ε, ατζέντα για την ΕΠΑ. Ε, τα κράτη-μέλη περιόρισαν τις φιλοδοξίες της Ένωσης στον τομέα αυτό και στην ουσία περιορίστηκε στην ε, πολιτική, στις πολιτικές δυνατότητες. Εγώ χαίρομαι που δεν συζητήθηκε το θέμα της ΕΠΑ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, διότι ήταν άσχετο θέμα. Η ΕΠΑ είναι επικάλυψη, επικάλυψη και καταστροφή. η απάντηση του ΝΑΤΟ στην κρίση που αντιμετωπίζουμε πώς στήθεται, Εγώ θεωρώ ότι είναι επιτυχημένη, αλλά πώς πλαισιώνεται. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Κώστερ. Ένα από τα προβλήματα είναι η δημόσια υποστήριξη και για στρατιωτική εμπλοκή και τις ε, στρατιωτικές δυνάμεις συνολικά το, έχει σκεφτεί κάπω καλύτερα το ΝΑΤΟ πώς μπορεί να ενισχύσει την υποστήριξη της κοινή γνώμης στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Μπορείτε να πείτε επίση και δύο λόγια για το τι γίνεται με το Συμβούλιο ΝΑΤΟ Ρωσία. Εγώ αν, κατάλαβα, κατάλαβα, έχω κατάλαβα καλά έχει παγώσει τελείω, αλλά πείτε μας δύο λόγια. Επίσης, ποια είναι η διαδικασία ανάπτυξη μια νέα στρατηγική στρατιωτική στρατηγική στρατηγικής του ΝΑΤΟ που θα αντικατοπτρίζει την επαναζωτικοποίηση της συμμαχίας. Κύριε Μαυρομιχάλη, η ρήτρα αλληλεγγύης είναι κάτι χρήσιμο εν δυνάμει για την Ένωση. Πάντα να βρίσκουμε χρήσιμο πράγματα καλό είναι και ο τομέας αυτός είναι ενδυνάμει ένα τομέας όπου θα μπορούσε να γίνει κάτι χρήσιμο, αλλά με, περι, με παραξενεύει γιατί το θέμα αυτό έχει να κάνει με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Είπατε ότι υπάρχει και εξωτερική και εσωτερική δράση, αλλά ο στόχος κατά βάση είναι εσωτερική αλληλεγγύη. Δηλαδή ένα κράτος μέλος ή περισσότερα ε, βοηθούν άλλα κράτη-μέλη. Σε περίπτωση μιας ε, πολιτικού χαρακτήρα καταστροφής. Και αναρωτιέμαι, πόσες, χρησιμο, πόσες φορές έγινε επίκληση αυτή τη ρήτας αλληλεγγύης μετά από την θέση της συνθήκη. Ευχαριστώ. Ο κύριος, η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Πρώτες μου ερωτήσεις απευθύνονται στον ε, κύριο Κώστερ στην ε, σύνοδο του ΝΑΤΟ στην ε, Ουαλία. Υπήρξε κάποιο σχέδιο δράσης που συζητήθηκε χωρίς να δημοσιευθεί. Η πρόσβαση που έχουμε στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αλλά σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε από τα μέσα ενημέρωσης είναι πως υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο είναι μέρος ενός ε, γενικότερου σχεδίου άμεσης ανταπόκρισης του ΝΑΤΟ. Αλλά ποιο είναι το εύρος ε, εφαρμογής αυτού του σχεδίου. Ακούγονται διάφορα νούμερα, διάφορες ε, χιλιάδες, αλλά ακριβώς τι γίνεται με αυτό. Έπειτα, τα επιμέρους μέτρα, για παράδειγμα, είναι σε στρατιωτικές ε, βάσεις. Αυτή η κορφή του δόρατος που αναφέρατε και πιο πριν, η ε, παγιοποίηση της ε, αμυντικής μας τάσης απέναντι στη Ρωσία. ποια είναι τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί για αποκλιμάκωση. Τι έχει γίνει ακριβώς. Και μία ακόμα ερώτηση για τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, κύριε Μαυρομιχάλη. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Βαν Όρτεν. Ο κύριος Βαν Όρτεν, έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, ρώτησε ε, τι έχει να κάνει η, Ευρωπαϊκή Αμερική Υπηρεσία με τις ε, κρίσεις, με τις εσωτερικές ε, κρίσεις. Διότι ασχολούνται και με στρατιωτικά ζητήματα. να πω ότι στα πλαίσια της ε, κρίσης έχουν δημιουργηθεί πολιτικές δυνατότητες. Και ποια η σχέση τους και η αναλογία τους με τις ε, στρατιωτικές δυνατότητες. Μας αναφέρατε ορισμένα σενάρια, για παράδειγμα, τα οποία αφορούν τις ε, ανθρώπινες καταστροφές. Θα μπορούσατε ίσως να μας ε, εξηγήσετε τι εννοείτε εσείς με τον όρο ανθρώπινες καταστροφές. Και πώς ακριβώς ε, γίνονται αντιληπτές αυτές οι ανθρώπινες καταστροφές. Γιατί το φάσμα είναι ευρύ και θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει και τις ε, μαζικές απεργίες, για παράδειγμα, ως μια τέτοια ανθρώπινη καταστροφή. Ε, μπορείτε να μας αποκλείσετε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπινων καταστροφών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μποντήλ Σεμπάγιος. Eh, eh, Ευχαριστώ. Κατάγομαι από μια χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και ε, ο, ο, ο λαός της Σουηδίας δεν τάσεται υπέρ μιας ένταξης της χώρα στο ΝΑΤΟ. Βέβαια, Έχουμε συνεργασία με άλλες σκανδιναβικές χώρες και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργασία σε θέματα άμυνας και μάλιστα έχουμε μία προετοιμασία για αμυντικά θέματα. Έχουμε συστήσει μία κοινοβουλευτική ομάδα που απαρτίζεται από βουλευτές που συνέρχονται τακτικά και εξετάζουν την κατάσταση ασφάλειας της Σουηδίας. Μάλιστα πρόσφατα συνεδρίασε αρκετές φορές η ομάδα αυτή και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η μεγαλύτερη απειλή για τη Σουηδία και το λαό της είναι ε, η κλιματική αλλαγή. Οι αλλαγές στο περιβάλλον. Αυτές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές ε, για την ασφάλεια, ε, οι σημαντικότερες προκλήσεις της ασφάλειας της Σουηδίας, οι κλιματικές αλλαγές. Βέβαια, μιλήσαμε για κάποια μετρά διαβεβαίωσης δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης που επικρατεί, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να σκεφτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η απειλή που προέρχεται από τις κλιματικές αλλαγές. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μείζον απειλή για τον πλανήτη. Και το θέμα φυσικά του πετρελαίου, το θέμα του φυσικού αερίου έχει κάποιες, δημιουργεί κάποιες απειλές. Αλλά σε όλο τον κόσμο έχουμε τόσες εμπόλεμες σειράξεις ε, και τόσα προβλήματα εξαιτία του πετρελαίου, εξαιτία της ε, μάχης ε, για τις πρώτες ύλε για τους φυσικούς πόρους. Γιατί δεν λαμβάνονται αυτά υπόψη στη συζήτηση για την πολιτική ασφάλεια, γιατί ξεχνάμε τόσο σημαντικά θέματα στην πολιτική ασφάλεια. Μιλήσαμε για τη ρήτρα αλληλεγγύης και τις ανθρωπογενείς καταστροφές. Έχω μια ερώτηση λοιπόν σχετική. Μήπως το θέμα αυτό θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε στη ρήτρα αλληλεγγύης. Μπορεί να ακούγεται λίγο παρατραβηγμένο, αλλά γιατί να μην το, γιατί να μην το διερευνήσουμε. Ο κόσμος Βοτόφσκι. Παρακαλώ, δεν σημείωσα καλά το όνομά σας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν θα σας κρύψω ότι είμαι ελάχιστα ικανοποιημένος. Όχι μόνο από τη σημερινή συζήτηση, αλλά και από προηγούμενες συζητήσεις. Γιατί έχω, τη έχω συνέστηση ότι έχουμε δύο παράλληλες πορείες. Έχουμε αφενός μια μεγάλη υψηλή πολιτική παιδεία των ε, καλεσμένων μας και μεγάλη διακριτικότητα σε ό,τι αφορά την ε, αποκάλυψη σημαντικών πληροφοριών. Ε, πού οφείλεται αυτό. Από οφείλεται στην έλλειψη γνώσης, στην έλλειψη σημαντικών πληροφοριών που μας ενδιαφέρουν. Γιατί δεν λαμβάνουμε τις πληροφορίες. Ή οφείλεται κάτι τέτοιο στην κατάσταση που επικρατεί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι στην προηγούμενη συζήτηση που έγινε πριν από μισή ώρα, τις πιο σημαντικές ερωτήσεις τις έθεσε ο κύριος Μάρεκ Γιούρεκ. Και δυστυχώς έμειναν αναπάντητες οι ερωτήσεις του κύριου Γιούρεκ. Αν λοιπόν δεν είστε ε, ε, έτοιμη, κυρία Πρόεδρε, να ζητήσετε απάντηση των, στις ερωτήσεις αυτές. Πώς θα σταθούν οι υπόλοιποι που αισθάνονται ανήμποροι απέναντι στην κοινή γνώμη που θέτει ερωτήσεις και μένουν απάντητες. Έχετε κάποιες ερωτήσεις συγκεκριμένες, ε, κύριε Ευρωβουλευτά. Οι ερωτήσεις μου αφορούν δύο θέματα. Υπάρχ, έχουμε γνώσεις, έχουμε πληροφορίες και γνώσεις για να απαντήσουμε αποτελεσματικά σε πολιτικές ή άλλες κρίσεις και είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες γιατί πολύ αμφιβάλλω. Δεύτερον, πολύ συχνά στις, ε, στα θέματα πολιτικής και άμυνας το πιο σημαντικό πράγμα είναι η γνώση γιατί Μιλήσαμε για τη δημιουργία ραντάρ, για τη δημιουργία συστήματος, πληροφορίες, ε, συστήματος πληροφοριών, ε, που ενισχύουν την κατάσταση της ασφάλειας. Δεδομένων των απειλών είμαστε ικανοί να αντιδράσουμε αποτελεσματικά με βάση τις γνώσεις μας και τις πληροφορίες μας. Τώρα, τι έγινε με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία. Δεν θεωρώ ότι ήταν επιτυχημένη αυτή η Σύνοδο Κορυφή. Έγιναν βέβαια τεράστιε προσπάθειε, πάσχησαν πολύ για να μην θεωρηθεί παταγώδη αποτυχία, αλλά επιτυχία δεν ήταν. Επίσης, η μη πρόσκληση της Ρωσίας ήταν επιτυχία. Αυτό είναι προφανές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έγινε κάτι καλό στην Ουαλία επειδή οι Ηνωμένε Πολιτείε χαρακτήρισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στρατηγικός εταίρος. Αυτό είναι για μας προφανές εδώ και πολλά χρόνια. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει τι, συνέβη, τι σημαντικό συνέβη στην Ουαλία, ώστε σύντομα να βελτιώσουμε την κατάσταση ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την ασφάλεια με την ευρία έννοια. και την ασφάλεια προς Ανατολάς. Πολύ σημαντικό είναι να ενισχύσουμε φυσικά την οικονομική ισχύ της Ευρώπης. Και η ασφάλεια της οικονομίας ε, της Ευρώπης ε, στηρίζεται και στην αμυντική πολιτική την δημιουργία ασφαλούς κλίματος για τους οικονομικούς φορείς. Αυτό θα πρέπει να το φροντίσουμε. Και δυστυχώς δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε εξασφαλίσει τέτοια προστασία. Ευχαριστώ πολύ, κύριο κύριος Τσάρλ Στάνο. Um, Σύντομη ερώτηση, πρόεδρε, σε συνέχεια του κύριου Βανόντεν. Προ ε, προς τον κύριο Μαυρομιχάλη πάντα να τον πιέσω. Έχετε συγκεκριμένα στατιστικά για το πότε για το κατά πόσον η ρήτρα αλληλεγγύης χρησιμοποιήθηκε για οποιαδήποτε μορφή είτε και πά είτε επά. Σας είπαν αν έγινε επίκληση. Αυτό έγινε για εσωτερικούς λόγους σε περίπτωση πλημμυρών ή άλλων ε, εθνικών καταστροφών, τρομοκρατίας, αλλά ε, ποια διάσταση και πά έχει προκύψει ποτέ, αν έχει προκύψει σε συνεργασία με τις συνθήκες. Η κύριε Άννα Γκόμες. Συνεχίζει κάποιος. Α. Υποστηρίζω απόλυτα αυτά που είπε ο στρατηγός για την σημασία της ανάγκης η Ένωση να αναδιαθρώσει την στρατηγική της ώστε να υλοποιήσει τον διάλογο με τον ΝΑΤΟ και να είναι πιο αποτελεσματική στο διάλογο αυτό. Ιδίως με τις απειλές που αντιμετωπίζουμε τώρα. Και αυτός είναι ένας άλλος τρόπος να αυξήσουμε την υποστήριξη της κοινή γνώμης για την ευρωπαϊκή άμυνα και παρεμπιπτόντως και για το ΝΑΤΟ. Έχω έρθει από ένα σεμινάριο για τους πυρηνικούς, βιοχημικούς ε, και λοιπούς κινδύνους, χειροβιπή κινδύνους. Ε, έχει γίνει κατανοητό πόσο προβληματική είναι η σημερινή κατάσταση με τον κατακαιρματισμό των προσπαθειών των χωρών της Ένωσης, ιδίως στο επίπεδο της διάγνωσης της, της, ε, και της προπαρασκευής. Εν ώψη των ανθρωπογενών καταστροφών που μπορούν να προκύψουν π.χ. από την κατάσταση στην Ουκρανία κάτι σε έναν πυρηνικό σταθμό ή από κρίσιμες υποδομές που είναι αντικείμενο αυτών των λεγόμενων ξένων μαχητών με υλικό που είναι εύκολα στα χέρια τους ή με πιθανούς ε, με τη χρήση όπλων με βιολογικό υλικό ή και όχι όπλων, ε, ε, ε, βιολογικού υλικού π.χ. του έμπολα. Εν ώψη των απειλών αυτών, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Καστάλντο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα με πολύ προσοχή και αρκετό ενδιαφέρον την παρέμβαση του κύριου Κουερμό και συγγνώμη αν προφέρω λάθος το επώνυμό σας. Είπατε, και το υπογραμμίζω αυτό, όταν αναφέρετε τις προτεραιότητες ε, μετά τη σύνοδο στην Ουαλία, ότι οι ΙΠΑ είναι αποφασισμένες να επιδιώξουν τους δικούς τους στρατηγικούς στόχους αλλού στον κόσμο. Εγώ θα ξεκινούσα από το σημείο αυτό για να υπογραμμίσω μια βασική αντίφαση που διαπιστώνεται συχνά ότι δεν είναι δεδομένο ότι τα συμφέροντα, οι προτεραιότητε δε της Ευρωπαϊκής είναι οι ίδιε πάντα με αυτές του ΝΑΤΟ. Και αυτό δημιουργεί κάτι άλλο που υπογραμμίσατε, την απουσία πραγματικής στρατηγικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίω δε την απουσία βούλησης πολλών κρατών της Ευρώπης να εξισορροπήσουν πραγματικά τις σχέσεις μεταξύ ΙΠΑ και Ένωσης στο εσωτερικό της συμμαχίας και για πολιτικούς λόγους. Κατά την άποψή μου, αυτό το βλέπουμε δραματικά εκεί όπου η Ευρώπη παίζει την αξιοπιστία της πραγματικά. Πιο κοντά μας. Μεσόγειο, για παράδειγμα, που, είναι, που φλέγεται απόλυτα. Λιβύη, Συρία, πριν από λίγο το ανθρωπιστικό δράμα της Γάζας μέχρι πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, ρωτώ με ποιο πώς συγκεκριμένα στην άπο, κατά την άποψή σας θα έπρεπε να προχωρήσουμε στη διαπραγμάτευση αυτής της συμφωνίας ασφάλειας και άνημινας μεταξύ Ένωσης και ΝΑΤΟ για να ξεπεράσουμε τον καματιγραμματισμό που αναφέρεται και να καταστήσουμε την Ένωση δρόντα παράγοντα πρώτης, ε, ε, βασικό παράγοντα στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Κύριε Κώστερ, μιλήσατε για σενάρια επιστροφής στον ψυχρό πόλεμο στην παρέμβασή σας. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η Ένωση δεν είναι ανεξάρτητη ενεργειακά, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης που είναι η μαζική επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ. Έχει κλείσει ο κατάλογος τώρα και προτού ζητήσω από τους εκλεκτούς καλεσμένους μας να απαντήσουν στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Θα ήθελα να απαντήσω στον Πολωνό συναδελφό μου. Ο στρατηγός Πατρίκ Τεροσχέ δήλωσε πρόθυμος για συνεργασία με την υποεπιτροπή μας για την ασφάλεια και την άμυνα. Μάλιστα, εγώ τον παρακάλεσα να συντομεύσει στην απάντησή του, γιατί η, η συζήτηση ήταν συναρπαστική, πολύ ζωντανή, έλαβαν μέρος πολλοί ομιλητές, τέθηκαν... τέθηκε πληθώρα ερωτήσεων και έτσι δεν ε, είχαμε χρόνο ε, για διεξοδικές απαντήσεις. Πάντως, ε, ο στρατηγός δήλωσε πρόθυμος για περαιτέρω συνεργασία και μάλιστα θα στείλει και γραπτές απαντήσεις σε μερικές ερωτήσεις. Και Όντως, μερικές ερωτήσεις έμειναν αναπάντητες, αλλά υποσχέθηκε ότι στις ερωτήσεις που δεν πρόλαβε να απαντήσει θα στείλει γραπτός απαντήσεις, τουλάχιστον στους συντονιστές ή στα μέλη που έθεσαν τις ερωτήσεις. Αυτά ήθελα να πω στον συνάδελφο και να δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας, ξεκινώντας από τον κύριο Πόστρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους ευρωβουλευτές για τα σχόλια και τις ερωτήσεις τους. Ας τα πάρω λοιπόν από την αρχή, θα προσπαθήσω να απαντήσω ένα προς ένα. Κύριε Γκάλερ, σχετικά με το αν οι νεότερες εξελίξεις θα ενισχύσουν την εφαρμογή και θα μπουν τα σχέδια αυτά στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια που βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αποστασιοποιηθεί κτλ. Δεν συμφωνώ κατά ανάγκη ε, με το ότι βρίσκονται στη σωστή θέση όλα αυτά τα στοιχεία. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δίνουν την ε, προσοχή του σε άλλα στρατηγικά σημεία στον κόσμο. Έχει γίνει συζήτηση τα τελευταία χρόνια για την ε, θέση που έχει η Ασία στις προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ πιστεύω πως οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ναι ε, στρέφουν την προσοχή τους και αλλού στον κόσμο, αυτό όμως ε, δεν μειώνει την προσοχή τους προς την Ευρώπη. Διότι αυτό που είδαμε εμείς στην Σύνοδο είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μια έντονη παρουσία στην Ευρώπη και είναι έτοιμε να συνδράμουν αν αυτό του ζητηθεί. Όσον αφορά την προσεχή μερίσια διάταξη τη ε, Συνόδου του ΝΑΤΟ, μπορώ να πω ότι μετά από τις ε, συζητήσεις που είχα σήμερα το πρωί, οι συνθήκες ε, μας οδηγούν αναπόφευκτα σε έναν καταμερισμό της εργασίας στο είναι πάρα πολύ σημαντικό η διάσκεψη κορυφής να έχει, η περσινή να έχει και συνέχεια την επόμενη χρονιά, διότι έτσι θα καθοριστούν απόλυτα οι προτεραιότητες της Ένωσης. Και αν συνδυάσετε τη δική μου παρουσίαση με εκείνη του κυρίου Μαυρομιχάλη, είναι σαφές το πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και εάν είναι σε θέση και σε ετοιμότητα να δώσει αποτελέσματα. Φυσικά, τα προβλήματα που αντιμετωπίσουμε είναι και θεσμικά. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εσείς οι πολιτικοί έχετε την δυνατότητα να το αλλάξετε αυτό. Δεν μπορεί να γίνει μέσω της γραφειοκρατίας αλλαγή. Κύριε Πάσκου, έχει συζητηθεί αυτό το επίπεδο εξουσίας και φυσικά θα βρίσκεται και αυτό στον διακανονισμό των ε, αρμοδιοτήτων που θα έχει αυτή η υψηλή ομάδα δράσης, η ομάδα δράσης υψηλής ετοιμότητας. Μιλάμε φυσικά για πάρα πολύ υψηλή ετοιμότητα και αυτό φυσικά προϋποθέτει και μια ε, ισχυρή εξουσία στο, κατά τον ψυχρό πόλεμο υπήρχε ένα αντίστοιχο κέντρο ελέγχου και επιχειρήσεων. Έχει συζητηθεί να αναπτυχθεί κάτι αντίστοιχο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορώ να σας πω πού θα οδηγήσουν ε, αυτά, αυτές οι εργασίες, όμως ναι, είναι μέρος αυτού του διακανονισμού. Τώρα, όσο για την άμυνα των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, αυτή είναι μια ερώτηση που θα αφήσω τους υπόλοιπου καλεσμένου να την απαντήσουν. Όμως, να σας πω ότι τα τα, οι χώρε που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ ε, είναι ευπρόσδεκτε να γίνουν. Κύριε Βανόρντεν. εάν υπάρχει έλλειψη στήριξη του κοινού. Ε, να σας πω ότι ο κύριος Πούτιν μας βοηθά πάρα πολύ να την αποκτήσουμε αυτή την ε, στήριξη από το κοινό. Μία στήριξη που θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε δυνατότητες και να αναπτύξουμε επίσης οι επιχειρήσεις, να αυξήσουμε τις αμυντικές εδαπάνες, να κάνουμε δηλαδή πράγματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να γίνουν πριν από 5 ή 10 χρόνια. Σίγουρα υπάρχει έλλειψη στήριξη από το κοινό σε ορισμένου τομεί, όμω πιστεύω πω ε, πάμε προ τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά το... την σχέση ΝΑΤΟ-Ρωσία, έχουμε αναστείλει την ε, συνεργασία σε υπουργικό επίπεδο, διατηρούμε όμω επαφέ σε επίπεδο πρεσβειών. Το Συμβούλιο δεν. Ε, δεν έχει πεθάνει, όμως είναι σε κόμμα θα έλεγα αυτή την εποχή. Και δεν ξέρω αν θα ξυπνήσει αυτό ο ασθενή που βρίσκεται σε κόμμα, όμω πιστεύω πω είναι προ το συμφέρον μα να κρατήσουμε ανοιχτού διάβλου επικοινωνία έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα στο μέλλον να ε, βελτιώσουμε τον διάλογο με την Ρωσία. Η Ρωσία τα τελευταία 20 χρόνια αναδείχθηκε σε πάρα πολύ σημαντικό εταίρο και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο κύριος Πούτιν απομακρύνεται από αυτό, όμως ελπίζουμε να αντιστραφεί η κατάσταση. Και εδώ απαντώ ταυτόχρονα και στην ε, ερώτηση της κυρίας Λέζιν για την ε, αποκλιμάκωση. Εμείς προσπαθούμε να στείλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα προς τη Μόσχα, πως είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και πως η απάντησή μας θα είναι αναλογική και πολύ καλά ζυγιασμένη. Και φυσικά εμείς δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση κλιμάκωση. Έχουμε όμως μία ευθύνη και η ευθύνη μας είναι η ασφάλεια των ε, μελών μας. Και αυτό φυσικά είναι κάτι που έχει κόστος και το ΝΑΤΟ ήταν σαφές προς αυτό. Και αν δείτε τι γίνεται από την άλλη πλευρά της ε, κλιμάκωσης, ε, είναι κάτι που δεν βρίσκεται δυστυχώς στο χέρι μας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις προκλήσεις της Μόσχας. Στόχος μας και πρόθεσή μας όμως σίγουρα δεν είναι η κλιμάκωση. Όπως είπατε, το σχέδιο αυτό του ΝΑΤΟ δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Η βάση μας δεν είναι πέντε κράτη, αλλά έξι, να σας πω. Και να σας πω ότι τα στρατιωτικά μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ είναι απόρριτα. Γι' αυτό δεν έχουμε την ελευθερία να συζητήσουμε μαζί σας όλες τις λεπτομέρειες του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Ωστόσο, η δήλωση που δημοσιεύτηκε μετά την ε, Σύνοδο μπορεί να σας δώσει πολλές απαντήσεις. Αν τη διαβάσετε θα δείτε ποια συστατικά στοιχεία θα αποτελούν το σχέδιο αυτό. Φυσικά το, το σχέδιο θα περιλαμβάνει περίπου 15.000 ε, στρατιώτες ως ε, στα πλαίσια της ομάδας άμεσης αντιμετώπισης και να σας πω επίσης πώς συνεχίζονται οι εξελίξεις για την ανάπτυξη του σχεδίου. Δεν μπορώ λοιπόν ακριβώς να σας πω ε, τι έκταση θα λάβει και πόσο θα είναι το εύρος του. Προσπαθούμε όμως να δώσουμε μορφή, ιδιαίτερα στη, στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα για τις ακριβείς τοποθεσίες όπου θα τοποθετηθούν αυτά τα στρατεύματα. Μπορώ όμως να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες ε, βάσεις ανεφοδιασμού, αν θέλετε, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ε, στρατεύματα και να, ε, σε περίπτωση ανάγκης και να καταφυγούν σε αυτές πάρα πολύ γρήγορα. Ε, να σας πω ότι υπάρχουν κάποια κεντρικά στην ε, Πολωνία, στα βορειοανατολικά. Δεν θα μπορέσω όμως να σας δώσω δυστυχώς περισσότερες λεπτομέρειες. Διότι αυτές, όπως σας είπα, είναι εν μέρη απόρριτες και εν μέρη ακόμα εξελίσσονται και αναπτύσσονται. Ο κύριος Ντρογεύσκη, αν διάβασα καλά το όνομά σας. Είπατε πως η σύνοδος δεν ήταν επιτυχής. Πιστεύω πως ε, ο πρόεδρός σας θα διαφωνήσει, διότι επέστρεψε από τη σύνοδο με ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον πολωνικό λαό ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται εκεί για εκείνους και πως η άμυνα της Πολωνίας είναι εξίσου σημαντική με την άμυνα των υπόλοιπων 27 κρατών μελών. και πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κάνουν ό,τι μπορούν για να υλοποιηθεί και να πάρει σάρκα και οστά αυτή η στήριξη. Και με ρωτήσατε πώς έχει βελτιωθεί η ασφάλεια από την σύνοδο μέχρι τώρα. Καταρχάς πιστεύω πως η σύνοδος δημιούργησε ένα μεγάλο αίσθημα ενότητας και κατανόησης πως συμμετέχουμε όλοι σε αυτό το project και πως πρέπει όλοι να συνδράμουμε σε εκείνους που αισθάνονται απειλή, που αισθάνονται, όχι απαραίτητα που υφίστανται. Υπάρχουν ήδη κάποια μέτρα που έχουν ληφθεί όσον αφορά την εναερία στην όμευση, όσον αφορά τις δυνάμεις στη θάλασσα και στην ξηρά. Ή ε, ορισμένα συστήματα ασφαλείας. Μπορείτε να δείτε επίσης τις λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ. Και πιστεύω, ναι, λοιπόν, πως έχει αυξηθεί και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αίσθημα ασφάλειας που έχουν οι πολίτες. Και θα υπάρξουν και επόμενα μέτρα που θα είναι περισσότερο διαρθρωτικού χαρακτήρα και θα αλλάξουν τη δομή του ΝΑΤΟ προς ε, μια πιο οριστική μορφή. Και θα αυξήσουν φυσικά και αυτά τα διαρθρωτικά μέτρα, την ασφάλεια. Έχουμε τον αμυντικό σχεδιασμό, τη λεπτομερέστατο σχεδιασμό, σχεδιασμό για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και δεν θα εστιάσουμε το μόνο στους ε, ανατολικούς μας συμμάχους αλλά και στις απειλές που θα έρθουν από τη Μέση Ανατολή, από το Ιράν, από τη Βόρεια Αφρική, το Ισλαμικό κράτος που αναπτύσσεται στο Ιράκ και τη Συρία. Η Σύνοδος λοιπόν πιστεύω ότι δημιούργησε και αύξησε την ασφάλεια των συμμάχων μας. Η ερώτηση του κύριου Κοστάλλου πιστεύω πως απευθύνθηκε περισσότερο στους ε, στον συνάδελφό μου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ε, ψυχρός πόλεμος, φυσικά και δεν είναι πρόθεσή μας να επαναληφθεί κάτι τέτοιο και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, που συμβαίνει και η απάντησή μας σε αυτό, έχει κάποια χαρακτηριστικά ψυχρού πολέμου. Δεν πιστεύουμε όμως ότι αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να πάμε και να οδηγηθούμε σε τέτοια είδους αντιπαράθεση παράθεση με τη Ρωσία. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποτρέψουμε αυτό. Και ιδιαίτερα και ως προς τις δυνατότητες που έχουμε, είμαστε σε πολύ διαφορετικό στάδιο από τη Ρωσία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρομιχάλης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να συμπτύξω τις ερωτήσεις που μου απευθύνατε και να δώσω σύντομες και περιστατωμένες απαντήσεις. Πολλοί ρωτήθηκαν αν η ΕΕΔΑ έχει, μπορεί να επηρεάσει τη ρήτρα αλληλεγγύης και πώς μπορεί να συμβάλλει στα θέματα αυτά. Φαίνεται ότι δεν ήμουν αρκετά σαφή στην προηγούμενη παρουσίασή μου, αλλά που δεν εννοούσα ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση διαδραματίζει κεντρικό ή αποκλειστικό ρόλο στην επίκληση της ρήτρας αλληλεγγύης. Η ρήτρα ελεγγύης ε, έχει στόχο την αντιμετώπιση κρίσεων στο έδαφος ε, των κρατών μελών, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τη ρήτρα αυτή, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται, συνενώνουν ε, τις προσπάθειες και την πραγματογνωμοσύνη τους προκειμένου να βοηθήσουν μια χώρα που επλήγει από τρομοκρατική επίθεση, θεομηνία ή ανθρωπογενή καταστροφή. Σας είπα ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης της ε, ρήτρα ε, ασφάλειας, ε, το κέντρο ανταπόκρισης σε κατεπίγουσες καταστάσεις θα έχει τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο. Αυτό το κέντρο θα είναι το σημείο επαφής. Εγώ σας παρουσίασα το ρόλο της ΕΙΕΔ και κυρίως ε, το ρόλο του τμήματός μου που είναι σημείο επαφής ε, σε θέματα αυτά και σας παρουσίασα τη δική μας συμβολή σε περίπτωση κρίσης ε, που δίνει λαβή για επίκληση της ρήτρα αλληλεγγύης και σε περίπτωση που έχει η κρίση αυτή και κάποια εξωτερική πτυχή. Για παράδειγμα, τρομοκρατική επίθεση στην επικράτεια μιας χώρας μέλους που σχεδιάστηκε στην αλλοδαπή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο εξωτερικό, κάτι που είναι πολύ πιθανό. Μπορεί για τα θέματα αυτά να έχουμε διαβαθμισμένες εμπιστευτικές πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αρκετοί ευρωβουλευτές διαρωτήθηκαν πόσο συχνά γίνεται επίκληση της ρήτρας αλληλεγγύης. Σας είπα ότι η ρήτρα ελεγγύης αποτελεί μια καινοτομία της συνθήκης της Λισαβόνας και μια κοινή πρόταση της ΥΠΑΤΗ εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποβάλλεται στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο έλαβε τη σχετική απόφαση στις 24 Ιουνίου του 2014. Πρόκειται για μια πολύ πρόσφατη απόφαση. Είχε μόνο τρίμηνη διάρκεια και στη διάρκεια του τριμήνου αυτού δεν έχει γίνει ακόμη επίκληση της ρήτρας ελληνικής και θα εξέφραζε και την προσωπική ευχή να μην γίνει ποτέ επίκληση της. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει ενεργοποιηθεί ούτε μία φορά η ρήτρα ελληνικής μέσα στη σύντομη διάρκεια ύπαρξής της, το τρίμηνο αυτό. Σας εξήγησα α, τις διαδικασίες. Είπαμε, πολλοί μίλησαν για τις χρονοβόρες διαδικασίες και την επαχθή γενικώ κινητοποίηση του μηχανισμού. Έχετε δίκιο, αλλά χρησιμοποιούμε και το IPCR, τις σχετικές διατάξεις ε, για την ολοκληρωμένη ανταπόκριση σε περίπτωση κρίσης. Πρόκειται για μια πλατφόρμα πληροφορικής ε, που μας επιτρέπει την ε, οργάνωση συνεδριάσεων και τηλεδιασκέψεων, ώστε να μπορέσουν τα κρατημέλη να μας στείλουν τις πληροφορίες τους ε, και τη συμβολή τους ε, σε θέματα πολιτικής προστασίας. Ε, αν κάποιος έστειλε αεροπλάνο με ιατρικές υπηρεσίες ή σκηνές ή κουβέρτες. Κάθε κράτος μπορεί να μας κοινοποιήσει τη συμβολή του, τη συνεισφορά του και Συγκεντρώνοντας αυτές τις πληροφορίες ε, μπορούμε και εμείς να δράσουμε στα πλαίσια φυσικά των αρμοδιοτήτων μας. Ρωτήσατε αν είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αλληλεγγύη σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εις βάρος κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι όμως και κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Όχι, δεν είναι αυτός ο ρόλος της ρήτρας αλληλεγγύης. Υπάρχει όμως άλλος μηχανισμός, άλλη διάταξη της συνθήκης, το άρθρο 42 παράγραφος 7, που προβλέπει ότι σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης ε, κατά κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το καθήκον να συνδράμουν το πλήγαν κράτος με βάση το άρθρο 51 και το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Και οι διατάξεις και του ΝΑΤΟ παραπέμπουν ε, και μάλιστα το ίδιο άρθρο παραπέμπει και σε κάποιες ρυθμίσεις του ΝΑΤΟ. Στόχος του άρθρου αυτού είναι να προβλέψει τέτοιο δεχόμενο. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε μια στρατιωτική επίθεση ως ανθρωπογενή καταστροφή. Οπότε απαντώ αρνητικά στη σχετική πρόταση ενό Ευρωβουλευτή. Τι είναι ανθρωπογενής καταστροφή. Μία καταστροφή που οφείλεται σε ανθρώπινο ε, λάθο ή σε ανθρώπινη ε, επιρροή. Ένα βιομηχανικό ατύχημα. Θυμάστε το Σοβέζο ή το ατύχημα του Μποπάλ στην Ινδία. Βέβαια δεν μπορούμε να εργοποιήσουμε τη δική μας ρήτρα αλληλεγγύης για την Ινδία, αλλά είχαμε και στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοιου είδους βιομηχανικά ατυχήματα. Οι κλιματικές αλλαγές ενδεχομένως θα μπορούσαν να προκαλέσουν συχνότερες θεομηνίες και άρα να οδηγήσουν σε επίκληση της ρήτρα αλληλεγγύης, αλλά οι κλιματικές αλλαγές από μόνες τους δεν συνιστούν ούτε θεομηνία ούτε ανθρωπογενή καταστροφή. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν τρομοκρατική επίθεση αναφέρθηκαν και άλλα προβλήματα και κρίσεις ε, πολύ εύστοχες ε, ερωτήσεις για τον ιό έμπολα για παράδειγμα. Αλλά η ρήτρα αλληλεγγύης ε, είναι ένα βήμα στο δρόμο του στενότερου συντονισμού των κρατών μελών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων προκειμένου να αντιμετωπιστούν μείζονες κρίσεις παρούσες ή μελλοντικές. Και χρειάζεται καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερη ολοκλήρωση και συνεργασία των επιχειρήσεών μας και το, του δυναμικού μας των επιστημόνων, της πολιτικής προστασίας, ακόμη και των στρατιωτικών δυνάμεων, γιατί μερικές φορές και ο στρατός συνδράμει σε περίπτωση μεγάλης θεομηνίας. Έτσι, θετώντας αυτή την ολοκληρωμένη τη σφαιρική προσέγγιση, που βρίσκεται στο επίκεντρο όλων μας των προσπαθειών, έχουμε και πιο αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων. Σας ευχαριστώ. Ο στρατηγός Γκομό. Με ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο, διότι πολλά ήδη αναφέρθηκαν. Κάποια εξωτερικά γεγονότα που αυξάνουν την επίγνωση της ανάγκης ευρωπαϊκής άμυνας και άμυνας γενικότερα. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι, εκπλή, δεν το ότι η ΕΠΑ δημιουργήθηκε την εποχή της Ιουγκοσλαβίας, του πολέμου στα Βαλκάνια. Η πρώτη φάση της ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας που ήταν το τι δεν είχε γίνει στο Ιράκ. Δηλαδή υπήρχαν πολιτικές και στατικές συμπτώσεις σε κάθε περίπτωση. Δυστυχώς, σε θέματα ασφάλειας άμυνας, σε γενικά στρατιωτικά, εάν υπάρχει κίνηση, η κίνηση αυτή γίνεται από εξωτερικά γεγονότα που σταδιακά κινητοποιούν κάποιες, κάποιο ενδιαφέρον και κάποια περαιτέρω κίνηση βλέπω ότι όλο και περισσότερο υπάρχει το θέμα της επίγνωσης. Να απαντήσω και σε μια άλλη ερώτηση. Δεν εδώ ο κύριος Βαρνόντεν, αλλά στην τελευταία σύνοδο κορυφής είπε ότι δεν ήταν επιτυχία. Εγώ νομίζω ότι ήταν, σε πολλούς τομείς. Να σας δώσω παραδείγματα. Η Επιτροπή μπαίνει μέσα κτλ. Αλλά το βασικό στοιχείο της ε, επιτυχίας της Συνόδου το Δεκέμβριο είναι ότι εν τέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινήσαμε με μια διαδικασία σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Και εσείς ζώντας εδώ σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ξέρετε τι σημασία έχει μια διαδικασία, μια εξέλιξη. Αυτό είναι σημαντικό. Θα διαφωνήσω λοιπόν με τον κύριο Βαν η ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας είναι εξαιρετικά σημαντική, ουσιαστική, ουσιαστική και ξανά ουσιαστική για την Ευρώπη. Για το πώς να αντιδρούμε γρήγορα και το ότι οι διαδικασίες που ακολουθούμε είναι κάπως βραβείες. Δεν ξέρω αν σας εκπλήσει αλλά εγώ ως στρατιωτικός σας έλεγα ότι οι διαδικασίες είναι εκεί για να μας βοηθούν. Οι στρατιωτικοί που ακολουθούν τις διαδικασίες, μόνο όμως τις διαδικασίες, χάνουν. Ε, καλό είναι να υπάρχουν διαδικασίες, αλλά μην ξεχνάμε και την πραγματικότητα των γεγονότων. Μία ερώτηση τώρα για, στην ερώτηση που θέσατε για το αν όντως η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια εμπλέκονται όλο και περισσότερο, η απάντηση είναι ναι. Τώρα για την ρήτρα αλληλεγγύης η απάντηση είναι όχι μορφής προέλευσης αλλά καθηκόντων. Σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τώρα δουλειές αστυνομίας δεν είναι πια δουλειά τη αστυνομία, δεν μπορούν να γίνουν από την αστυνομία, αλλά χρειάζονται και την παρέμβαση του, των στρατιωτικών. Στην ε, χώρα μου υπάρχει η δυνατότητα παρέμβαση του στρατού σε περίπτωση που η πολιτική, ε, η πολιτική δύναμη, δηλαδή η αστυνομία, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εάν σε μια χώρα υπάρχει δήλωση της κυβέρνησης ότι κοιτάξτε η πολιτική προστασία μου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην συγκεκριμένη επίγουσα κατάσταση, χρειάζεται στρατιωτική παρέμβαση, θα πούμε όχι, νομίζω ότι η ρήτρα αλληλεγγύης επιβάλλει να κάνουμε κάτι τέτοιο. η κυρία Γκόμες έδωσε ένα πολύ καλό παράδειγμα όπου ε, μπορούν να βοηθήσουν οι πολιτικές και οι στρατιωτικές διαστάσεις της ρήτρας αλληλεγγύης. Οι κίνδυνοι χείρο VP μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφή πολύ γρήγορα και εκεί πρέπει να κινητοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη θέσή μας. Οπότε και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη σχέση ΝΑΤΟ και ΕΠΑ. Μια προκλητική πρόταση θα μπορούσε να είναι η εξή. Στο ΝΑΤΟ υπάρχουν πολύ καλής ποιότητας μόνιμο στρατηγείο που προχρηματοδοτείται από χώρες της Ευρώπης που επανδρώνουν Ευρωπαίοι στρατιωτικοί. Τη μέρα που θα χρειαστεί, χρειαστεί ένα τέτοιο στρατηγείο για διαχείριση κρίσης, δεν ξέρουμε αν θα εμφανιστεί. Άρα πρέπει να το βελτιώσουμε. Ένα παράδειγμα μεταξύ Βελγίου και Ολλανδία. Υπάρχει ένα στρατηγείο για το ναυτικό. Αν μετάσχουν και οι δύο χώρες σε μία δράση, κανένα πρόβλημα. Αλλά αν η μία χώρα πει ναι και η άλλη όχι, έχουμε ένα στρατηγείο που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η διοίκηση μπορεί να είναι εθνική, αλλά τα στρατηγεία θα παραμείνουν. Αν κάποιες χώρες πούν τώρα ότι θέλω να, δεν θέλω να κρατήσω το προσωπικό μου ε, στο στρατηγείο μπορεί να το αποσύρει. Αυτό είχε γίνει και με την αποχώρηση της Γαλλίας. Η βοήθεια μπορεί να δοθεί μόνο σε αυτούς που θεωρούν ότι ανεξάρτητα από το που είναι το στρατηγείο, το, προσωπικό μου μένει εκεί. Αυτό είναι η συνέργεια μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει ότι δεν σπαταλούμε ικανότητες. Μη δείτε το στρατηγικό πλαίσιο, το στρατηγικό στρατηγείο, δηλαδή το, το ουσιαστικό στρατηγείο, το περιβάλλον εκεί είναι πολύ καλό. Τελειώνω εδώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαντλήσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς ε, καλεσμένους στο πάνελ μας για αυτό το σημείο που εξετάσαμε στην ημερήσια διάταξη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συνεδρίαση της ε, Επιτροπής αυτής. Θα συνεχίσουμε στις 3 το μεσημέρι, όπου θα ασχοληθούμε με το επόμενο σημείο, δηλαδή την ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Συρία, το Ιράκ και το Ισλαμικό κράτος. η οποία θα γίνει μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το σημείο. Ah au revoir.